Ε, ε, επίκληση της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Η ομάδα μου ήταν υπέρ της έκθεσης. Παρακαλώ την Κομισιόν, τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να την ε, διαβάσει και να την μελετήσει και ακόμα και αν σε αυτό το σημείο δεν ισχύει η συναπόφαση, παρόλα αυτά τα θεμητά ε, τις θεμητές απόψεις του Κοινοβουλίου θα πρέπει να τις λάβει υπόψη και να απαντήσει στην τελευταία ερώτηση επί της ουσίας που θέσαμε στην τελευταία έκθεση για τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, αν ο βασικός κανονισμός είναι ο 1203 και μήπω θα πρέπει αυτός να τύχει επεξεργασίας βραχυπρόθεσμα ούτως ώστε οι μεσαίες επιχειρήσεις να διαφοροποιούνται από τι μεγάλες όταν πρόκειται για την επιβολή προστήμων. Είναι σημαντικό λοιπόν να ε, έχουμε μια αποτελεσματική και επικοδομητική απάντηση, όχι γενικόλογη. Ευχαριστώ, κατά τα άλλα ε, συμφωνώ. Ευχαριστώ κύριε Σουάμπ. Η κυρία Βάιλερ για τους σοσιαλιστές. Παρακαλώ. Α, ακούσαμε Βάιλερ. Ακούσαμε Βάιλερ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κρίνο Μπουσό για την έκθεσή του. Ήμουν στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, γι' αυτό καθυστέρησα λίγο. Για το σημείο 5 που αφορά το τομέα των φαρμάκων, ε, νομίζω ότι είναι πραγματικά μεγάλε οι ανησυχίε και πολύ σωστά τονίζει αυτά που τονίζει για το φαρμακευτικό τομέα. Γιατί θα πρέπει να δώσουμε στο τομέα αυτό τη σημασία που το αρμόζει. Για την ενέργεια, ίσω και σε αυτό, στο 4 δηλαδή, θα έπρεπε να αναφέρουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών στην ε, εσωτερική αγορά. Αν υπάρχει αλλαγή δηλαδή φορέα παρόχου ε, τι μπορεί να γίνει. Δεν έχει να κάνει δηλαδή το θέμα μόνο με τις τιμές, αλλά και η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και στην περίπτωση αλλαγής ε, παρόχου. Και βέβαια θα συνεργαστώ με τον συζητητή για βελτίωση του κειμένου. Ευχαριστούμε. Συμφωνώ με τον κύριο Σβάμπ που λέει να ρωτήσω με την Κομισιόν για τις συνέπειες που και τα συμπεράσματα που συνάγει από τις εκθέσεις είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί α, κα, ε, τι νόημα έχει κάθε χρόνο να κάνουμε την έκθεση και να είναι μια ρουτίνα. Πολύ σημαντικό λοιπόν να ερωτηθεί κατά τα άλλα. Συμφωνώ με τις προτεραιότητες του εισηγητή. Η ενέργεια είναι πολύ σημαντικό θέμα, το πιστεύω και εγώ και ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα έχουν υψηλή, υψηλό βαθμό συγκέντρωσης πολλέ ε, πολλές μέλη. Αυτό έχει επιπτώσει και για τους καταναλωτές. Επίσης ε, θα πρέπει να δούμε και την ε, λειτουργία των δικτύων. Να δούμε δηλαδή τι πολιτική ακολουθείται σε αυτό το τομέα, τι προτάσεις υποβάλλονται σε αυτό το τομέα. Αυτή είναι η δική μου παρατήρηση. Τώρα το μίλησα ως σκιώδης για τους πράσινους. Και τώρα ο κύριος Μπίλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα με τη διερμηνία. Χαίρομαι που βλέπω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άρχισε να δουλεύει νωρίτερα ε, φέτος. Υπάρχει πρόβλημα. Στα γερμανικά υπάρχει πρόβλημα. Ναι, ναι, υπάρχει πρόβλημα εδώ με την ε, τεχνική μας γιατί δεν ακούμε τη μετάφραση. Ε, τα γερμανικά δεν τα καταλαβαίνουμε. Γαλλικά δεν ακούγονται καθόλου. Yeah. better. Okay. Okay. We have to wait. Czy mam powtórzyć? Do I have to repeat what I just said? Uh, um, να επαναλάβω, να επαναλάβετε. Παρακαλώ. Ε, για να δούμε και όλα, αρχίστε για να δούμε και αν λειτουργεί το σύστημα. Μιλήστε στα πολωνικά και να δούμε αν λειτουργεί. Λίγα λόγια να πείτε. Ωραία. Τώρα είναι εντάξει. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι θερμά τον κύριο Μπούζοη για την προετοιμασία της έκθεσης. Χαίρομαι πολύ διότι τώρα θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την έκθεση ταχύτερα από ό,τι πέρσι. Νομίζω ότι με μια φωνή πρέπει να μιλήσουμε. Νομίζω ότι έχουμε πολύ λίγο χρόνο Χαίρομαι διότι ο κύριος Μπούζοη επικεντρώθηκε στους δύο τομείς ενέργεια 2000, γιατί το 2009 ήταν ένα έτος κατά το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, ενέκριναν το πακέτο για την ενέργεια και επ' αυτού του θέματος ε, αφιερώνεται πολύ χώρο στο έγγραφο της Κομισιόν. Η δε επιλογή του φαρμακευτικού τομέα επίσης είναι πολύ επιτυχής. Πολλά πρέπει να γίνουν. Θέλω να ευχαριστήσω το, θερμά τον κύριο Μπούσοη που μίλησε και για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Γιατί στο βαθμό που δεν υπάρχει δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στην ολοκλήρωση της κοινή αγοράς. Εδώ μία αντίφαση μόνο βλέπω στο σημείο 3 συγκεκριμένα όπου πρόκειται για την συλλογική αρρωγή των θυμάνων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαλντίνη. Όχι, δεν ζητεί το λόγο. κύριος Ζουβέν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του. Ε, δύο-τρεις ε, παρατηρήσεις θέλω να κάνω ε, ενδεχομένως εν είδη τροπολογιών. Πρώτο ζήτημα, ε, την φαρμακευτική βιομηχανία ε, για την οποία έγινε ήδη λόγος η έννοια του ε, διπλώματος ευρεσιτεχνίας που καθυστερεί την είσοδο στην αγορά ε, γενικών ε, γαλλικών φαρμάκων βεβαίως είναι μια ιδέα σωστή αλλά στην ουσία μας ενδιαφέρει περισσότερο η κατάχρηση των ευρεσιτεχνιών ε, όλο αυτό, το, ζήτημα για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ε, βεβαίως είναι ε, καλή ιδέα να βρεθεί ένα τρόπος έτσι ώστε εάν κατατεθεί η ευρεσιτεχνία σε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε να θεωρείται κατατεθειμένη σε όλες τις χώρες ε, πολύ σημαντικό. Ε, και ένα τελευταίο σημείο όσον αφορά τις ε, συλλογικές προσφυγές. Έγινε λόγος πολύ για αυτό το θέμα. Το ζήτημα είναι να ξέρουμε εάν οι πολίτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν συλλογική ε, ε, να κάνουν έτοιμα συλλογική αποζημίωσης ε, εάν μπορούν να το κάνουν σε εθελούσια βάση ή αν θα γίνεται με κάποιο είδος αυτοματισμού και αν θα πρέπει απλώς να προσυπογράφουν ένα opting in. Ο κύριος Μάιερ και μετά η Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το δίκαιο του ανταγωνισμού είναι κομμάτι της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, σημαντικότατο κομμάτι της μάλιστα και χρειαζόμαστε ένα νομικό πλαίσιο σε όλες τις ε, ανθρώπινες σχέσεις και στην οικονομία της αγοράς. Αυτό είναι θεμελιώδες ε, ζήτημα. Ε, υπάρχει το δίκαιο για τα καρτέλ, ένα άλλο κομμάτι αφορά τη διαφήμιση και τώρα θέλουμε, και αυτό είναι το μοναδικό μας καθήκον και μέλημα, να απελευθερώσουμε την εσωτερική αγορά μέσα σε ένα πλαίσιο ένομης τάξης όμως. Γιατί πάντα θα πρέπει να ισχύει αυτό για τη συμβίωση των ε, λαών 27 κρατών μελών. Τώρα, πόση ελευθερία θα ε, προβλέψω, τι περιορισμούς θα θεσμοθετήσω. Η ελευθερία υπάρχει στη διαφήμιση και τα όρια είναι εκεί που αρχίζει η κατάχρηση. Πολύ σωστά επικεντρώνεται σε καταχρηστικές πρακτικές ο εισηγητής. Καταχρηστικές πρακτικές μιας επιχείρησης που παρουσιάζεται ως καταναλωτή και μπορεί να βλάψει ευάλωτες ομάδες, ε, ανηλίκους κλπ. Το ζήτημα είναι, δεν μπορούμε να είμαστε λίγο πιο γενικό, γενικοί ε, στην προσέγγιση μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια γενικότερη φύσεως απόφασης, γιατί τίνομαι σε μεμονωμένους, ε, σε μεμονωμένους τομείς δικαίου, δικαίου καταναλωτών κλπ, να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Ο καθένας που έχει μια ιδέα υποβάλλει μια τροπολογία και πάμε σε 600, από 600 μέχρι 2.000 τροπολογίες, που είναι ανόητο πολλές φορές. Θα πρέπει να επικεντρωνόμεθα πιο πολύ σε βασικές γραμμές και αρχές και μετά, ναι, πιστεύω ότι είναι σωστό ότι το θέμα της ενέργειας, όπως λέει ο εισηγητής, ναι, να το δούμε. Αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφεύγουμε τις 1.600 τροπολογίες, να δουλεύουμε πιο καθαρά, πιο στοχευμένα, να συζητούμε και να ε, εξετάζουμε γενικές αρχές και όχι ε, συγκεκριμένες υποθέσεις. Αυτό είναι δουλειά των δικαστηρίων. Απευθύνω έκκληση λοιπόν. Αυτό το θέμα της ελευθερίας της εσωτερικής αγοράς και των περιορισμών στα πλαίσια μιας ένομης τάξης και πλαισίου. Ναι, αυτό πρέπει να το επεξεργαστούμε για να προστατεύσουμε τους καταναλωτές, αλλά θέλουμε και τις επιχειρήσεις να προστατεύουμε με μεγαλύτερη καθαρότητα στις θέσεις μας, με μεγαλύτερη σαφήνεια. Πιστεύω ότι πολλές φορές ε, ε, υπησερχόμεθα σε υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες ε, και αυτό δεν είναι καλό. Ούτε έχει νόημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπούμε στις λεπτομέρειες των 27 κρατών μελών με τις διαφορές τους και τις παραδόσεις τους τις διαφορετικές. Ε, οι καταχρηστικές πρακτικές είναι στο στόχαστρό μας. Δεν μπορεί να μπαίνουμε και να ρυθμίζουμε την κάθε άνθιπο λεπτομέρεια. Θα ήταν λάθος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μάιερ. Η Κομισιόν, η κυρία Μπρούμς από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίζει το προσχέδιο έκθεσης του εισηγητού Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και θεωρεί ότι το κείμενο ε, αναφέρεται σε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία της πολιτικής ε, ανταγωνισμού. Ε, και βεβαίως θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον ε, εισηγητή για τα εύσημα τα οποία απονέμει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την ε, κρίση που ξεκίνησε πέρσι. Θέλουμε να προχωρήσουν οι χρηματοοικονομικές αλλαγές όσο γίνεται πιο εύκολα. Αλλά βεβαίως, όπως είπε και ο Επίτροπος Αλμούνια προημερών, δεν θα μπορέσουμε να άρουμε τους ε, περιορισμούς ε, και τις ε, προϋποθέσεις μέχρι το, τις αρχές του 2012 και τότε θα μπορέσουμε να πιέσουμε και τις τράπεζες έτσι ώστε να άρουν τις προϋποθέσεις τις οποίες έχουν και έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα των κρατικών βοηθειών. Ε, πρώτον, ε, είναι ε, γεγονός ότι εμείς έχουμε την Γενική Διεύθυνση η οποία ασχολείται με την προστασία των καταναλωτών. Επίσης έχουμε το Consumer Liaison, αυτήν την έννοια του συνδέσμου καταναλωτών που ασχολείται με την πρόθεση των ειδικών προβλημάτων. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό μοντέλο συλλογικής αρρωγής, Βεβαίως ε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υπάρξει ένα πρώτο προσχέδιο το οποίο θα ε, μπει σε διαβούλευση από τον Νοέμβριο μέχρι τέλη Φεβρουαρίου. Ο Αντιπρόεδρος ε, Αλμούνια στο Συμβούλιο Ανταγωνισμού την προηγούμενη εβδομάδα ανήγγειλε ότι όταν το Συμβούλιο εγκρίνει το πλαίσιο τότε θα περιληφθούν και διαφορετικά πεδία εφαρμογής όπως ας πούμε περιβαλλοντικός ανταγωνισμό ανταγωνισμός, προστασία καταναλωτών κτλ. Επίσης, ε, έχει ε, στο δεύτερο μισό του 2011 συμφωνηθεί ε, να υπάρξει και ανακοίνωση σχετικά με το μοντέλο συλλογικής αλλαγής θυμάτων παραβίασης νομοθεσίας. Ε, και ε, θα προωθηθεί με τρόπο ώστε να υπάρξει ένα πρότυπο για όλους και μία κατάσταση για όλους αλλά βεβαίως σε σεβασμό των εθνικών νομικών ε, υποβάθρων. Αυτό είναι, αυτή είναι η βάση των αποφάσεων. Πρώτο βέβαια θέμα στη σειρά είναι ε, το ε, πλαίσιο συζητήσεων το οποίο και διαβουλεύσεων που θα διαρκέσει από τον Νοέμβριο μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπόσχεται ότι και δεσμεύεται ότι όλες οι, όλα τα σημεία τα οποία θα αφορούν τον ανταγωνισμό ε, θα εγκριθούν με τρόπο ώστε να προστατεύεται και ε, το δίκαιο των καταναλωτών. Όσον αφορά τώρα την εσωτερική αγορά ενέργεια. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει τις ανησυχίε που εκφράζει ε, και ο εισηγητής και οι σκιώδες εισηγητές ε, πρέπει να σας πω όμως ότι ήδη το 2009 και το ε, παρόν, ε, το τρέχον έτος έχουμε ήδη ξεκινήσει δράσεις κατά αυτή την έννοια. Όσον αφορά τον φαρμακευτικό τομέα, ήδη εμείς έχουμε ξεκινήσει δράσεις και ερχόμαστε σε επαφή με εκπροσώπους του κλάδου έτσι ώστε να καταλάβουμε καλύτερα τα προβλήματα. Όσον αφορά την, το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα και την λύση διαφωνιών ε, όσον αφορά ε, το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Εύρεση Τεχνίας. Ε, υπάρχουν ανακοινώσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά αυτή την έννοια και αυτές θα πρέπει να αποτελέσουν βάση για περαιτέρω συζητήσεις. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές και όλους τους άλλους συναδέλφους οι οποίοι εξέφρασαν μια πολύ θετική άποψη σε σχέση με τις ιδέες που προτείνω στο σχέδιο γνωμοδότησής μου. Προσβλέπω λοιπόν και στις τροπολογίες που θα λάβω για να βελτιωθεί και το κείμενο. Συμφωνώ πλήρως με τον κύριο Σβάπ, με την κυρία Στάιλερ, με εσά κυρία Πρόεδρε, καθώς και με τον κύριο Μπίλαν και τις ιδέες που εκφράσατε όλοι. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία που έλαβε να ξεκινήσει τη συζήτηση για την οδηγία, για την αποζημίωση σε ό,τι αφορά τον κύριο Ζουβέν Συμφωνώ και εγώ ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις ε, καταχρήσεις ό,τι αφορά τα φάρμακα κοινόχρηση της ονομασίας. Και για το opt-in που είπατε για τη συλλογικέ συλλογικές προσφυγές. Αν μπορείτε να μου υποβάλλετε τροπολογίες ε, και για τη βελτίωση του κειμένου, με αυτά χαρά να τις ε, συμπεριλάβω στο τελικό μου κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. 28 Δεκάτου, 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Οπότε ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και πάμε στο επόμενο. Α, ο κύριος Ζουβά. Ο κύριος Ζουβά. Είναι η έκθεση του κυρίου Ζουβάν τώρα που θα συζητηθεί. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Ζητώ συγγνώμη. Ε, έβλεπα λίγο τις ε, σημειώσεις μου. Πρώτα απ' όλα, πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας, η οποία γνώρισε μια σχετική <laughs> επιτυχία, γιατί έχουμε 130-140 τροπολογίες. Θα ήθελα εξ αρχής, κυρία Πρόεδρε, ε, να σας πω ότι η έκθεση αυτή ε, που ονομάζεται Αντίκτυπος Διαφήμισης Συμπεριφορά των Καταναλωτών να ασχοληθεί πολύ με το διαδίκτυο, με το ίντερνετ, γιατί αυτός, ο, γιατί ε, στην ουσία η παραδοσιακή διαφήμιση ε, ήδη αποτελεί αντικείμενο πολλών νομοθεσιών. Οι νέες μορφές μετάδοσης του διαφημιστικού μηνύματος πρέπει να μας ενδιαφέρει περισσότερο. Το πρώτο τμήμα της έκθεσης υπενθυμίζει ε, τα θετικά στοιχεία της ε, διαφήμισης, τα ωφέλη της διαφήμισης. Δεν θέλουμε ε, να με κανένα τρόπο να ρίξουμε στο πυρ το εξώτερο την διαφήμιση, αλλά θέλουμε να υπενθυμίσουμε και όλα τα άσχημα και όλες τις καταχρήσεις οι οποίες μπορούν να υπάρξουν. Επίσης, αναφερόμαστε στις νέες πρακτικές οι οποίες διοχετεύονται μέσω των νέων τεχνολογιών, οι οποίες θα πρέπει να ρυθμιστούν ε, ε, υπενθυμίζοντας πάντως ότι εμπιστευόμενοι τους ε, επαγγελματίες βλέπουμε ότι η αγορά της διαφήμισης αυτορυθμίζεται ικανοποιητικά και μέχρι ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχει βέβαια μια φιλοσοφική συζήτηση για την διαφήμιση που θα πρέπει να μας οδηγήσει όμως σε ορθολογικά ε, μέτρα και σε λογικές ε, διαστάσεις. Δουλέψαμε με επικοδομητικό νομίζω τρόπο με τους συναδέλφους νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα για ε, συμβιβαστικές τροπολογίες σε πολλά θέματα. Παραμένουν κάποια σκληρά σημεία τα οποία ενδεχομένως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα ας πούμε η πρακτική του opting που κατά την άποψή μου δεν είναι ε, δυνατή και θα δυσκολέψει την πλοήγηση στο ίντερνετ κατά την άποψή μου. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να επιλέξουμε το privacy ε, by design δηλαδή από την αρχή, από, την, το σχεδιασμό να υπάρξουν παράμετροι ασφάλειας, είναι ένα ε, ζήτημα το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο αλλά είναι ευρύ και ενδεχομένως ε, εδώ έχουμε πολλές αποκλίνουσες απόψεις. Αναφέρομαι στην προστασία ε, του ονόματος της μάρκας. Ξέρετε ότι ενώ ε, προστατεύονται οι μάρκες παρόλα αυτά γίνεται, πολλούνται μέσω διαφήμισης από πολλούς φορείς του ίντερνετ. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να βοηθήσουμε την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων γιατί αυτή είναι η υπεραξία μας. Επίσης όσον αφορά τα υνοπνευματόδη κάνω μια πρόταση μάλλον σκληρή κυρία Πρόεδρε. Ε, δηλαδή στην ουσία εγώ λέω ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρης απαγόρευσης ε, εξαιρουμένων κάποιων συγκεκριμένων ε, επαγγελματιών. Να υπάρξει λέω πλήρης απασχόληση διαφήμισης του εινοπνεύματος, γιατί είναι θέμα δημόσιας υγείας και ε, στο ίντερνετ μονάχα οι τοπικές αρχές, οι ε, αρχές του τουρισμού, το ε, γραφεία τουρισμού κατά τόπους και επαγγελματίες να μπορούν να κάνουν διαφημίσεις για υνοπνευματώδη στο διαδίκτυο. Αυτά είναι ε, τα τρία σκληρά κατά κάποιο τρόπο σημεία επί των οποίων μάλλον δεν θα υπάρξει συμφωνία. Στα υπόλοιπα νομίζω ότι τα πράγματα είναι αρκετά απλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, Ισκιώδης, ο κύριος ε, Παντσίρη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζουβάν ε, γιατί ε, παρουσίασε μια σειρά τροπολογιών που ενσωματώνουν ε, τις ε, παρατηρήσεις που είχαμε ε, υποβάλει και παρουσιάσει στην τελευταία συνάντηση της Ίνκο. Δεν θα επανέλθω λοιπόν σε αυτά. Υπάρχουν όμως ε, κάποια σημεία τα οποία δεν καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς και ελπίζω ότι από αυτόν θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποιες συμβαστικές λύσεις ε, μαζί με τον συνάδελφο ε, Γνώκα έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες και πρέπει να πω ότι ε, σε αυτές τις τροπολογίες υπάρχει κάποιο πρόβλημα ε, δηλαδή ε, στις τροπολογίες 2, 22, 18, 63, 49 λείπει το όνομά μου από το, ως συγγραφέα ε, των τροπολογιών παρακαλώ τη γραμματεία να το σημειώσει και να το διορθώσει μόνο στην ιταλική εκδοχή υπάρχουν λοιπόν κάποια σημεία ακόμα στην αιτιολογική σκέψη α θεωρούμε ότι θα πρέπει να διατυπωθεί με τρόπον ώστε να ε, διατυπώνεται ότι η διαφήμιση είναι σημαντικό στοιχείο του ανταγωνισμού, ε, μπορεί να αποτελέσει δυναμικό στοιχείο ε, της πρόθεσης των προϊόντων και άρα της πρόθεσης της αγοράς. Στο, στην αιτιολογική σκέψη ή e, αναφέρεται η, θα πρέπει να πούμε ότι ε, ναι μεν θα προστατεύεται η προσωπική ζωή ε, αλλά ότι από τη στιγμή που οι καταναλωτές δώσουν ε, την σύμφωνη γνώμη τους δεν θα υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την διαφήμιση. Όπως είπε και η συγητής προηγουμένως για θέματα, για στοιχεία μάλλον όπως είναι ή για αγαθά όπως είναι τα υνοπνευματόδη, όπως είναι τα τυχερά παιχνίδια, προϊόντα καπνού κτλ. Ε, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την, ε, ε, το ίντερνετ έτσι ώστε να αποφύγουμε τα προϊόντα απομίμησης αλλά και την, τον εθισμό σε ορισμένες περιπτώσεις. Επίσης, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια βασική νομοθεσία αλλά ταυτοχρόνως να έχουμε και εναρμονισμένη αντιμετώπιση του τομέα της ε, διαφήμισης. Αυτό στην παράγραφο 5. Στην παράγραφο 7 πιστεύουμε ότι ε, θα πρέπει να πούμε ότι η αυτορύθμιση του κλάδου δεν μπορεί να υποκαταστήσει ε, το νομικό πλαίσιο. Στην παράγραφο 11 πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει λόγος για την ανάγκη ύπαρξης εκστρατιών πληροφόρησης και στην παράγραφο 12 αναφέρεται ότι τα η θεματική των ε, διαφημίσεων που αποτελούν ε, ε, που πρέπει να απαγορευθούν συγγνώμη που έχουν περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό που ρυθμίζεται από τα νομικά πλαίσια θα πρέπει απλώς να απαγορευτούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο ο Σκιώδης για τους φιλελευθέρους. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη που άργησα, αλλά είχε σταματήσει το μετρό μεταξύ δύο σταθμών και είχα μπλοκαριστεί. Θέλω να συγχαρώ φυσικά τον συνάδελφο Ζιβά και για την έκθεσή του, αλλά και για το πολύ σημαντικό έργο το οποίο επιτελεί, ώστε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Βέβαια δεν άκουσα τι είπε πριν, ε, άκουσα μια περίληψη μόνο. Όπως και ο εισηγητής έτσι και εγώ νομίζω από την αρχή ότι πρέπει την έκθεση αυτή ε, να τη λάβουμε υπόψη μας, αντιλαμβάνοντας υπόψη το ότι γίνεται στο διαδίκτυο. Βλέπω και στο Κοινοβούλιο ότι έχουμε κείμενα που ενώ είναι πάρα πολύ ευραία, εκ πρώτη όψεω, ε, ουσιαστικά έχουν να κάνουν με ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Με κοιτάει ο Αντρέα. Βλέπω λοιπόν ε, και θέλω να του πω κιόλας ότι δεν το λέω μόνο για τη δική του έκθεση αυτό. Συμφωνώ με τα περισσότερα σχόλια του κυρίου Ζυβά, Όπως και ο κύριος Ζιβάτς και εγώ θεωρώ ότι ορισμένες από τις τροπολογίες ίσως να μην έχουν ως στόχο την ε, εξέβριση μιας ισορροπίας μεταξύ του στόχου της διαφήμισης ε, στην ευρωπαϊκή αγορά και της αποτροπής αρνητικών ε, αποτελεσμάτων. Ούτε πρέπει να σας πω ότι στην αρχή ήμουν και πεπισμένος πώς να το εκφράσω σε ό,τι αφορά παραδείγματο χάρη την προστασία του εμπορικού σήματο, δεν ήξερα ότι υπάρχουν αρπακτικοί, αν θέλετε, ε, καταναλωτέ οι οποίοι θα πήγαιναν να αγοράσουν προϊόντα χωρί να υπάρχει μια προστασία. Τέλο πάντων, δεν ξέρω ακριβώ τι γίνεται. Σίγουρα, αν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, η πνευματική ιδιοκτησία που δεν περιορίζεται σε αυτό, είναι και η βιομηχανική ιδιοκτησία. Είναι, ε, μιλάμε και για την οικονομική ανάπτυξη εδώ. Θα πρέπει λοιπόν να λαμβάνονται υπόψη αυτά τα θέματα. Κάτι που δεν είναι και τόσο απλό είναι το ζήτημα των πνευματοδών. Νομίζω αν κατάλαβα καλά θα ήθελες να το περιορίζουμε σε επαγγελματίε, γιατί υπάρχει ζήτημα δημόσια υγεία. Το καταλαβαίνω αυτό. Νομίζω ότι το αλκοόλ δεν είναι πολιτιστικό αγαθό. Ε, εγώ θα έλεγα ε, να συμφωνήσουμε με την αρχική μείωση. Γιατί θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη και το επιχείρημα που μπορεί να έχουν τα γραφεία τουρισμού. Εγώ προέρχομαι από μια περιφέρεια με πολύ σημαντική αμπελοϊνική παραγωγή. Εντάξει, αν βγάλουμε την περιφέρεια του Μπορντό που είναι στην περιφέρειά μου, ε, είναι σημαντική πρωτεύουσα πάντως το Μπορντό σε ό,τι αφορά την περιφέρεια αυτή. Ίσως γύρω από τα γραφεία τουρισμού θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Τώρα ε, δεν ξέρω ποια χαρακτήρα θα είχαν αυτές οι οργανώσεις εκεί, θα έπρεπε να το δούμε αν θα ήταν επαγγελματικέ Τώρα, ε, σε ό,τι αφορά τι τροπολογίε, κάποιοι συνάδελφοι από την ομάδα μου έχουν υποβάλει τροπολογίε, δεν του βλέπω όμω εδώ. Αλλά θα ήθελα να συζητήσουμε με λοιπόν, τον κύριο Ζιβά των προτέρων για να τα βρούμε αν θέλετε, αλλά του το εξήγησα ότι λόγω κάποιων κινητοποιήσεων ήταν και έκθεση δεν μπόρεσα να το κάνω, πάντως είμαι στη διάθεσή του. Μέχρι την ψηφοφορία στην Επιτροπή, μήπως μπορέσουμε και συμφιλώσουμε κάποιες απόψεις. Συγγνώμη, πατώ το λάθο κουμπί για το μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τούρνεν, για του πρασίνους. Ευχαριστώ, ευχαριστώ ε, πολύ, κυρία Ζουβάν, για την εξαιρετική δουλειά. Είναι εύκολο να είναι κανεί σκιώδη όταν έχουμε τόσο εξαιρετικό σημείο θετηρίας. Αυτό εισαγωγικά. Πολλέ τροπολογίες είναι όμοιες Κάποια πράγματα θα συζητήσουμε για το, για το ενόπνευμα για παράδειγμα και ορισμένα άλλα που είναι σημαντικά για μας τους πρασίνους που θα τα δείτε όταν διαβάσετε τις τροπολογίες. Καταρχήν η αναφορά στην οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές που πρέπει να τροποποιηθεί λιγάκι, να μπουν κάποιες αποχρώσεις, γιατί υπάρχουν δυσκολίες εισαγωγής της πλήρους εναρμόνισης. Υπάρχουν σχετικές ε, αποφάσεις του δικαστηρίου για την προστασία των καταναλωτών που ε, εξασφαλίστηκε σε ορισμένε χώρες, αλλά το θέμα είναι προβληματικό και αυτή η αναφορά θα πρέπει να ε, συμπληρωθεί και να αποτελέσει τμήμα της αξιολόγησης της οδηγίας από την Επιτροπή. Πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε, να δούμε αυτή η αρχή της πλήρους εναρμόνισης τι σημαίνει σε ένα τόσο ραγδαία μεταλλασσόμενο τομέα. Πρέπει να υπάρχει μεγάλη ευελιξία από τα κράτη-μέλη για να ακολουθούν αυτές τις νέες ε, εξελίξεις. Αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε και να ενημερώσουμε την Κομισιόν. Δεύτερον, η συζήτηση για τα ε, προσωπικά στοιχεία, privacy. Αυτό ε, το συμπληρώσαμε ως privacy by design, ως αρχή που θα πρέπει να ε, συνεχιστεί και ενδεχομένως θα μπορούσαμε να ε, κάνουμε λίγο πιο δυναμικό το κείμενο, το κείμενο για τα θέματα αυτά της ιδιωτικής προστασίας. Αυτά τα δύο από την πλευρά μας θέλαμε να τονίσουμε ως θέματα, κατά τα άλλα είναι πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Η κυρία Παντσέρη η μετάφραση του κειμένου στα Ιταλικά καθυστέρησε λιγάκι, ε, λήφθη υπόψη αυτό που είπατε, ε, θα το φροντίσουμε. Τα άλλα μέλη της Επιτροπής τώρα. Η κυρία Στάιλερ, καταρχήν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Νομίζω ότι ο αριθμός των τροπολογιών δείχνει το ενδιαφέρον που υπάρχει για την έκθεση. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για την ενίσχυση της διαφήμισης ε, για τα που στοχεύει τα παιδιά. Εσείς συμφωνείτε με αυτές τις τροπολογίες που ενισχύουν ε, και τονίζουν περισσότερο το θέμα. Επίσης για ε, την οδηγία θέμη των εμπορικών πρακτικών, στο αρχικό ψήφισμα γινόταν λόγος ε, για ανανέωση σε τακτική βάση. Καλύτερα είναι να πούμε σε αιτήσια βάση, να το προσδιορίσουμε. Θα ήθελα να μας πει τι σκέπτεται ο εισηγητής για όλες αυτές τις τροπολογίες για τα παιδιά. Μίλησε για το ενόπνευμα πώς θα τονίσουμε περισσότερο το θέμα και θα ε, βεβαιωθούμε ότι θα υπάρχει μια ενημέρωση σε αιτήσια βάση σχετικά με τις αθέμητες ε, εμπορικές πρακτικές. Ο κύριος Μάιερ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Ο Φιλίπ Ζουβά με ενθουσιασμό και επάρκεια ασχολήθηκε με το θέμα. Δεν τίθεται θέμα επ' αυτού. Οι διαφημίσεις είναι σημαντικό θέμα της καθημερινότητας, όπως και το Facebook πια. Όλοι σχεδόν είναι στο Facebook. Και βέβαια εκεί δεν υπάρχει προστασία δεδομένων όταν ε, ενταχθεί κανείς ε, σε ένα τέτοιο δίκτυο. Τι σημαίνει διαφήμιση. Μην τη δαιμονοποιούμε σημαίνει ότι πάμε να επηρεάσουμε κάποιον που θα δει τη διαφήμιση ή θα την ακούσει, ώστε να αλλάξει την αγοραστική του συμπεριφορά. Ε, ο επηρεασμό είναι το νόημα της διαφήμισης, οπότε δεν θα, το, δεν θα ασχοληθούμε με αυτό. Βέβαια, το θέμα είναι πάλι, όπως είπα και πριν, πότε αρχίζουν οι καταχρηστικές πρακτικές. Δεν είναι τίποτε περισσότερο. Όλα τα άλλα σωστά τα είπατε, προστασία της πνευματικής ε, ή διανοητικής ιδιοκτησίας. Υπάρχουν ορισμένοι ε, νόμοι, γι' αυτό υπάρχει το δίκαιο για τα σήματα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι τόσο καλό και θα πρέπει να τύχει κατεπηγόντως επεξεργασίας. Γιατί έχουμε μεγάλες μάρκες στη Mercedes, στην Siemens, στην ε, Γερμανία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά πηγαίνετε να αγοράσετε ένα προϊόν Siemens σε ένα κατάστημα. Δεν υπάρχει αυτό η διαφήμιση ε, επηρεάζει πολύ και βέβαια και άλλα ε, δίκαια επιμέρους θα έχουμε ε, επιμελώς ρυθμίσει στην Ευρώπη. Πάλι ξαναλέω αυτό που είπα. Μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Εγώ είμαι εντελώς αντίθετος. Δεν μπορεί να προβαίνουμε σε απαγορεύσεις σε όλους τους τομείς. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε όταν πρόκειται για ακραία θέματα. όταν δηλαδή υπάρχουν πολύ σοβαρές ε, ε, παρεμβάσεις αρνητικές για την υγεία, για την αγορά κλπ. Και γι' αυτό έχω κάνει τη σχετική τροπολογία μαζί με άλλους συναδέλφους ότι η διαφήμιση του ινοπνεύματος δεν θα πρέπει να απαγορεύεται όπως προτείνεται με τόση αυστηρότητα πάντα θα πρέπει να σκεπτόμεθα. Πρέπει να γίνει αυτό, γιατί ο στόχο μα είναι η ελευθερία της εσωτερικής αγοράς. Δεν θα κουράζομαι να το λέω αυτό. Η ελευθερία της εσωτερικής αγοράς είναι το σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολλά εμπόδια έχουμε καταργήσει και τώρα τα ξαναβάζουμε από την πίσω πόρτα. Προσοχή λοιπόν σε αυτά τα θέματα. Ε, υπάρχουν επίσης και περιφερειακές διαφορές πρέπει να διαφυλάξουμε κάποια επικουρικότητα εδώ και θα πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στα κράτη-μέλη ότι και εκείνα θεσπίζουν ε, σωστή νομοθεσία στην επικράτειά τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάντερ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ε, Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή για την πρόταση. Συμφωνώ επίσης με πολλούς από τους ομιλητές Συνήθως είμαι υπέρ των εθελοντικών συστημάτων. Εντάξει, μπορεί κάποιος να μπορεί να ουσιαστικά να τηρήσει την νομοθεσία, αλλά αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω εδώ και λείπει σχέτιση με το ποινικό δίκαιο για να υπάρχει επιβολή. Δηλαδή, αν εταιρείε ή άτομα παραβαίνουν, παραβιάζουν το, την νομοθεσία, να υπάρχει δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτό που βλέπω είναι ότι εισάγουμε νομοθεσία χωρίς όμως δυνατότητα επιβολής της τελικά. Είμαι λοιπόν υπέρ κάποιων εθελοντικών ε, συστημάτων και αν εισαγάγουμε κάποιες απαγορεύσεις στην νομοθεσία θέλω εγώ να δω να εισάγεται και η δυνατότητα επιβολής και ίσως ακόμη και επιβολή κυρώσεων πρόστιμων. Τουλάχιστον να είναι δυνατό να επιβληθούν πρόστιμο. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μακλάρκιν που ήρθε από την ECR. Θέλετε να μιλήσετε για την έκθεση Ζουβάν. Ή πρώτα να δώσουμε το λόγο στον ομιλητή. Α, τώρα θέλετε. Δεν θέλετε. Ο κύριος Ζουβάν. Και μετά η κυρία Λάρκιν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται όπως είπα και προηγουμένως ε, για έκθεση πρωτοβουλίας. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια ευκαιρία να υπενθυμίσουμε μεγάλες αρχές. Μεταξύ αυτών των αρχών λέμε ότι πρώτον η διαφήμιση είναι απαραίτητη για την οικονομική δραστηριότητα, δεύτερον ότι εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε την προσωπική ζωή, να προστατεύσουμε τα ευάλωτα άτομα, και κατηγορίες ατόμων και ότι όλα τα στοιχεία αυτά δεν αντιτίθενται το ένα στο άλλο και εμείς το καταδεικνύουμε ε, στην έκθεσή μας. Και στην ερώτηση πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες κύριε Μάγερ, εγώ λέω ότι ένας τρόπος λειτουργίας είναι να προτείνουμε ε, στοιχεία λεπτομέρειας έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Δεν σας κρύβω ότι σαν νέος βουλευτής, είμαι ένα χρόνο περίπου εδώ, βρίσκω ότι μερικές φορές ε, ότι οι εκθέσεις ε, πρωτοβουλίας είναι ε, έτσι λίγο ασκήσεις επιχάρτου και εγώ θα ήθελα πέρα από την άσκηση επιχάρτου να έχουμε και κάποιο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Συμφωνώ με τον κύριο Ροσφόρ. Πιστεύω ότι ότι σίγουρα είναι περίπλοκο θέμα και από αυτού δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, όμως πιστεύω ότι εδώ υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας. Είναι δύσκολο να πει κανεί ότι το ενόπνευμα είναι καλό για την υγεία. Μια γαλλική ομάδα πριν από μερικά χρόνια έκανε μια εργασία σύμφωνα με το οποίο το ε, ε, κρασί ήταν καλό για την υγεία. Αλλά τι να σας πω τώρα, εγώ δεν πείθεομαι τόσο εύκολα και ούτε για τον Μπορντό πιστεύω ότι το να πίνει κανείς Μπορντό κάνει καλό στην υγεία, ε, αλλά υπάρχουν και θέματα ε, πολιτισμικά τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να βρούμε ε, ε, σίγουρα μία λύση. Έχει δίκιο ο κύριο Ροσφόρ ότι θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στις υπηρεσίες τουρισμού και ενδεχομένως σε κάποιους παραγωγούς που συνδέονται ε, με το γραφείο του τουρισμού να τους δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν κάποια διαφήμιση για τα προϊόντα τους. Όσον αφορά την κυρία Στάιλερ, ε, κυρία Στάιλερ, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο το οποίο να μπορεί να προσαρμόζεται ε, καλύτερα στην παρούσα πραγματικότητα. Ίσως θα πρέπει εδώ να ρωτήσουμε και τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω όμως ότι μια ετήσια αναθεώρηση ε, είναι πολύ βαριά και μπορεί να μπλοκάρει το όλο σύστημα. Ενδεχομένως ε, θα πρέπει να ζητήσουμε αναθεώρηση οποτεδήποτε εμφανίζονται ε, νέες τεχνολογίες. Η Επιτροπή θα μας πει. Όσον αφορά τώρα τα άλλα στοιχεία, προστασία των παιδιών, των ευάλωτων ομάδων, βεβαίως θα πρέπει να εμφανίζονται τα στοιχεία αυτά στην έκθεση. Αλλά θα ήθελα η αναφορά να μην είναι επαναλαμβανόμενη μια και είναι ένα θέμα που μας, ένα ζήτημα που μας αφορά όλους, ε, θα μπορεί κανείς να βρει στοιχεία σχετικά σε διάφορα σημεία της έκθεσης. Εγώ θα ήθελα να έχουμε μια συνθετική ε, παρουσία. Δηλαδή να υπάρχει το, το θέμα αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά όχι κάθε δύο-τρεις γραμμές να το αναφέρουμε. Αυτά είναι τα σχόλια τα οποία ήθελα να κάνω. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανείς από την Κομισιόν σήμερα για να σας δώσει απαντήσεις. Κρίμα. Υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία θα λάβει χώρα 8 Νοεμβρίου για την έκθεση αυτή και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. Ε, κυρία Μακλάρκιν, έχετε το λόγο για την παρουσίαση της έκθεσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Η ανακοίνωση τη Επιτροπή για τη Μείωση των Ανισοτήτων στον τομέα τη υγεία εντοπίζει την ανάγκη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε διάφορου τομεί πολιτική ώστε να υπογραμμιστούν τα κοινωνικό και άλλα αίτια των ε, ανισοτήτων στον τομέα τη υγεία. Είναι ένα αχανέ ε, θέμα, ένα αχανή τομέα. Δεν μπορούμε φυσικά να το καλύψουμε πλήρω στην Επιτροπή μα. Ελπίζω όμω να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις και να το προσανατολίσουμε σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά, τη σκοπιά της εσωτερικής αγοράς. Προτάσεις δράσης της Κομισιόν στο μήνα αυτής περιλαμβάνουν τη βελτίωση της ανταλλαγής και συλλογής δεδομένων, βελτίωση των μηχανισμών για την μέτρηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ανισότητων στον τομέα της και στα κράτη-μέλη υποστήριξη των αρμόδιων εθνικών αρχών, ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμφάνιση των πολιτών να συμμετέχουν ε, στην ε, σχετική συζήτηση, ανάπτυξη και συνεργασία σε διάφορου τομεί πολιτική για την ανταπόκριση στι ανάγκε των πιο ευάλωτων ομάδων. Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει καμία συγκεκριμένη δράση σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά ή την πολιτική προστασία των καταναλωτών. Υπάρχει πάντως σαφή ε, θέση που θα πρέπει εμεί να υιοθετήσουμε από την πλευρά τη ε, εσωτερική αγορά για να εξασφαλίσουμε την εξάλληψη των ανισοτήτων στον τομέα τη υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θέλω να συζητήσουμε μαζί σήμερα. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα, την προσιτότητα των θεραπείων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την καταπολέμηση των ανισοτήτων στον τομέα τη υγεία. Στον τομέα, οι διαφορέ ε, στα φάρμακα μπορεί να, στις τιμές των φαρμάκων μπορεί να δημιουργήσει ε, πολλά προβλήματα. Υπάρχουν διατάξεις για την εναρμόνιση και σε ό,τι αφορά την αποζημίωση. ό Είναι η σχετική οδηγία για τη διαφάνεια. Βέβαια υπάρχουν κάποια άλλα μοντέλα τιμολόγηση ε, οθούμενα από την αγορά, τα οποία θα προσφέρουν πιο αποτελεσματικά. Επίση, ενημέρωση των ασθενών, κατά απομίμηση φαρμάκων, είναι και άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να τα εξετάσουμε. Και έχουμε συμβάλει με σχετικέ γνωμοδοτήσει ω ΣΥΜΚΟ. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι ανοιχτά στη δυνατότητα χορήγηση ευέλικτων αδειών κυκλοφορία φαρμάκων. Γιατί έτσι μόνο θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την έρευνα, τι επενδύσει και βέβαια την καινοτομία στον τομέα τη οικονομική περίθαλψη. Δεύτερον, για τη βελτίωση τη συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων σε επίπεδο κρατών μελών και Ευρωπαϊκή Ένωση θα μα δώσει ε, πολλά στοιχεία, ίσω και για τα υποκείμενα αίτια. Επίσης, ανταλλαγή τεχνικών καλών πρακτικών, ε, ανταλλαγή πληροφοριών για τα αποτελέσματα των ε, θεραπείων, ε, κακές πρακτικές ε, και επίσης συνεργασία με τις τοπικές αρχές που ξέρουν καλύτερα πού εντοπίζονται οι ανισότητες στον τομέα της υγείας. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι φορείς να μπορούν να συζητούν αυτά τα στήματα και νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει εδώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρίτον, σε ό,τι αφορά την διασυνοριακή υγεία, τη σχετική οδηγία και εδώ μπορούμε να επηρεάσουμε. Πρόκειται βέβαια για ένα ξεχωριστό νομοθέτημα που στόχο έχει να δημιουργήσει μια ενιαία αγορά για του ασθενεί. Αλλά μπορούμε να εξετάσουμε το πώ θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο των υπηρεσιών υγεία ε, τι ανισότητε. Μπορούμε να δούμε ότι και η ίδια γεωγραφική θέση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το επίπεδο ή την ποιότητα των υπηρεσιών που μπορεί να έχει ένα ασθενή. Ουσιαστικά είναι λαχείο. Δηλαδή, ακόμη και ασθενεί ε, στην ίδια περιοχή μπορεί να έχουν τελείως διαφορετική θεραπεία. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες και τις ανισορροπίες αυτές και να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα για αυτή τη διασυνοριακή υγεία, για αυτή μια σχετική διάταξη. Δεν θα πρέπει να βλέπουμε μόνο τη δημόσια υγεία, αλλά να έχουμε μια ευρύτερη προσέγγιση. Εμεί έχουμε εδώ σημαντικέ προτάσει στον τομέα τη επισήμανση των τροφίμων, την προστασία των καταναλωτών, τη διαφήμιση όπως και ο πίνακας επιδόσεων για τους καταναλωτές είναι επίσης πολύ σημαντικό για να εντοπιστούν ανισότητες. Προπαρασκευαστικές δράσεις στον τομέα επίσης ε, της σωματικής δραστηριότητας, του αθλητισμού μπορούν να βοηθήσουν κατά πολέμηση των ανισοτήτων. Και ίσω θα πρέπει όλε αυτέ οι διαφορετικέ πτυχέ να ενταχθούν στην έκθεση. Τέλο, το σημαντικότερο είναι ότι τις ανισότητες μπορούμε να τι αντιμετωπίσουμε αν προωθήσουμε την αμοιβαία αναγνώριση, δηλαδή αν προωθήσουμε την εφαρμογή τη οδηγία, για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Μήπω θα μπορούσε να υπάρχει ένα σύστημα για την αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων, να υπάρχει ένα σύστημα λογοδοσία και για τι μετακινήσει των εργαζομένων, καθώ και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών. Θα πρέπει επίση να διερευνήσουμε τι ε, διάφορε δοκιμάσει που υπάρχουν στα επαγγελματικά προσόντα μεταξύ κρατών μελών και να δούμε αν αυτό επηρεάζει ή όχι και τα προσόντα των ιατρών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σύστημα ε, πληροφοριών ή το σύστημα συναγερμού προειδοποίηση που θα μπορούσε να ενταχθεί το εξετάζει αυτή η Επιτροπή, όπως εξετάζει και το κατά πόσον θα μπορούσε η εντός ε, του χώρου εργασία ε, επιμόρφωση να βοηθήσει στη βελτίωση των μελλοντικών προσόντων. Όλες αυτές τις πτυχές μπορούμε και εμείς να τις διερευνήσουμε. Κάνοντας κεντρική πτυχή τη γνωμοδότησή μα ε, τα επαγγελματικά προσόντα. Οι ανισότητε λοιπόν στον τομέα τη υγεία είναι ένα σημαντικό βάρο για τα κράτη-μέλη αλλά και για το υγειονομικό σύστημα κάθε χώρα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 60 δι είναι απόλυτα παραγωγικότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των ανισοτήτων. Το Εθνικό Σύστημα υγεία πλήττεται και Βέβαια δεν μπορούμε να το εξετάσουμε στην γνωμοδότηση, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που δεν ισχύει μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και για όλα τα κράτη-μέλη. Βέβαια, δεν χρειάζεται να υπάρχει ξεχωριστό θεματολόγιο υγεία για να αντιμετωπιστούν οι ανισότητε. Θα πρέπει σε ευρύτερα και στην οικονομία και στα κοινωνικά θέματα να ληφθεί υπόψη η πτυχή αυτή. Για ανοιχτέ και ανταγωνιστικέ αγορέ, επίση, πρέπει να πω ότι αν υπάρχουν μπορούν να βοηθήσουν και μπορούν να βοηθήσουν και τα κράτη-μέλη να βρουν πιο ευέλικτες και αποτελεσματικέ λύσεις. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα ήθελα τώρα να ακούσω τους σκιώδεις και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπάστος παρακαλώ για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Μακλάρκιν για την πολύ ξεκάθαρη και στεναρή αυτή παρουσίαση. Θέλω να πω ότι η ανακοίνωση της Κομισιόν δημιουργεί ένα πλαίσιο ρεαλιστικό και αντικειμενικό για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκαθαρίζει το θέμα ε, με επικέντρωση στις σοβαρές ανισότητες ε, σε σχέση με κάποιους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπογραμμίζονται επίσης με τρία παράδειγμα ε, θνητότητα βρεφών κάτω του ενός έτους, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιοχές με πενταπλάσια βρεφική θνησιμότητα από τις σε άλλες και επίσης ε, Υπάρχει διαφορά 14 ετών στο προσδόκιμο ζωής μεταξύ περιοχών για τους άνδρες και υπάρχουν και πολλές διαφορές στην περίθαλψη. Αυτά τα παραδείγματα λοιπόν δείχνουν το πλαίσιο που θέτει η Κομισιόν και φαίνεται έτσι ότι χρειάζεται σαφής απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα αυτά. Η έκθεση θα καταρτιστεί Τώρα, όπως ξέρετε, η Κομισιόν θα ασχοληθεί με αυτά τα θέματα που θα χειριστεί η συγγήτρια Έντιτε Στρέλα και η συγγήτριά μας υπογράμμισε πολλά ζητήματα που την απασχολούν σε ό,τι αφορά τις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Το θέμα είναι ότι παρακολουθήσαμε εκ του σύνεγγις το έργο των εθνικών τόσο περιφερειακών όσο και τοπικών αρχών στον τομέα της υγείας. Το έργο τους είναι κέριο. Θα πρέπει να υπάρξει ανανέωση της εστίασης στους ίδιους τους πολίτες για να διασφαλίσουμε ότι και οι πολίτες θα προάγουν τα συμφέροντά τους και τα δικαιώματά τους για την υγεία. Πρέπει να επικεντρωθούμε στις ευάλωτες ομάδες, τους φτωχούς, τους άνεργους, τους ανάπηρους, τα παιδιά, τα βρέφη ειδικότερα. Οπότε αυτή η περίοδος που περνάει με τώρα στην Ευρώπη είναι μια περίοδος ανεργίας, ε, δημοσιονομικής, χρηματοοικονομικής κρίσης, κοινωνικής κρίσης, οπότε τώρα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ε, ισότητα των ευκαιριών. Επίσης έχουμε και πολλά παράδοξα φαινόμενα. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η περικοπή των δαπανών και η εφαρμογή μέτρων λιτότητας, περικοπές δημοσίων δαπανών από τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να λυθεί το πρόβλημα του ελλείμματος του προϋπολογισμού. Βέβαια, το λογικό αποτέλεσμα οποιασδήποτε αναθεώρησης των δαπανών είναι ότι τα ποσά που έχουν αφιερωθεί στην υγεία, στον προϋπολογισμό, θα περικοπούν. Αυτό είναι μια προσπάθεια αποτελεσματικότερης διαχείρισης που θα επηρεάσει όμως τους πόρους που διατίθενται για τις υπηρεσίες υγείας στα κράτη-μέλη. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το έχουμε ιδιαίτερα υπόψη μας κατά την ε, σύνταξη της έκθεσης. και την έκθεση της Έντιτε Στρέλα στην υπό αρμόδια επιτροπή. Αυτά για το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ομιλήτρια η κυρία ε, Βαρνιό για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που μας έδωσε τα μηνύματα για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κύμα της Επιτροπής πράγματι πολύ σωστά εντοπίζει τις ανισότητες στο τομέα της υγείας. Ε, τις έχουμε και εμείς πολύ σωστά εντοπίσει, όπως έχουμε εντοπίσει νομίζω και τις ευάλωτες ομάδες το των λεχθέντων, η ανισότητα στον τομέα της υγείας. Ε, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το αναπόφευκτο. Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και έχει επιπτώσεις σε όλες τις πολιτικές μας και στο επίπεδο της εσωτερικής αγοράς. Γι' αυτό δεν θα έπρεπε να νομίζουμε ότι αυτή η οικονομική κατάσταση τόσο δύσκολη ε, σε ό,τι αφορά την οικονομική, δαφική, τοπική συνοχή θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσχημα για να αλλάξουμε την πολιτική υγείας που εφαρμόζουμε. Οι ανισότητες στον τομέα της υγείας υπάρχουν. Η υγεία έχει κόστος, δεν ε, μπορούμε όμως ε, να μην την παράσχουμε. Δεν έχει τίμημα θα έλεγα. Υπάρχουν επίσης διαφορετικές ε, συνθήκες στα κράτη-μέλη, διαφέρει κατάσταση στην Ήπεθρο ε, σε σχέση με τα αστικά κέντρα, οπότε στην Ήπεθρο θα πρέπει κανείς να δει τις λεγόμενες ευαίσθητες περιοχές όπου υπάρχουν άστεγοι, υπάρχουν ε, μετανάστες και που είναι δύσκολο να τους εντοπίσει κανείς, μπορεί δύσκολα κανείς να δει ποιες είναι οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, ε, η κατάσταση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Έχουμε εντοπίσει πάντως δύο ομάδες τους νέους που μπορεί να έχουν κάποιες επικίνδυνες συμπεριφορές, μιλώ κυρίως για την αντιμετώπιση του αλκοολισμού. Όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό σήμερα ακόμα, και λιγότερο φτωχές. Και δεύτερον, ο γυράσκων πληθυσμός, ιδίως όταν ε, είναι και άστεγοι ή δεν έχουν κάποια προστασία. Σε όλες τις πολιτικές πρέπει να ενταχθεί η διάσταση, η συνδεγιορική πολιτική, η περιβαλλοντική, ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εργασία, για την ασφάλεια στην εργασία. Και εδώ μπορούμε να βελτιώσουμε για την καταπολέμηση, την πρόληψη των ανισοτήτων. Φυσικά και πρέπει να ενισχύσουμε τα ερευνητικά μας προγράμματα. Το, progress, το πρόγραμμα Progress πρέπει επίσης να συμβάλλει και αυτό στην καταπολέμηση των ανισοτήτων, αλλά αυτό που πρέπει να δούμε είναι το εξή. Εγώ θα ήθελα να σταθούμε στον ορισμό, σε ό,τι αφορά την υγεία, τον ορισμό που δίνει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, που λέει ότι η υγεία είναι μια κατάσταση φυσικής και πνευματικής ευεξίας και όχι μόνο η έλλειψη ε, ασθενειών, παθήσεων. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη και στην έκθεσή μας. Ολοκληρώνοντας, φυσικά, θα πω και δεν εξαρτάται από την Επιτροπή μας, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν προγράμματα πρόληψη στα σχολεία. Αυτό δεν εξαρτάται βέβαια από την Επιτροπή μα, Ωστόσο, αυτό το οποίο εξαρτάται από την Επιτροπή μα και ελπίζω να σημειώσουμε γρήγορα πρόοδο, θα έχουμε και μια συνάντηση σήμερα το απόγευμα, είναι η εναρμόνιση των επαγγελματικών προσόντων για όλου του επαγγελματίε του τομέα τη υγεία που ταξιδεύουν, που μετακινούνται και ιδίω θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ε, ε, απερίμωση και την έλλειψη γιατρών ε, στην Ήπεθρο θα πρέπει να άρουμε αυτή την νομική ασάφη που υπάρχει, αυτή την νομική αβεβαιότητα που ταλανίζει όλου του επαγγελματίε του τομέα τη υγεία. Ευχαριστώ και ελπίζω να συνεργαστούμε γιατί το θέμα είναι και πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για τους φιλελεύθερους, δεν είναι εδώ η κυρία Παρβάνοβα που είναι σκιώδη. ο κύριος Μπουζόη θα μιλήσει. Ναι, είναι η κυρία Παρβάνο Βασκιώδης, αλήθεια είναι αυτό, αλλά δεν μπόρεσε να έρθει. Θα παρουσιάσω κάποιες ιδέες. Καταρχήν, συγχαρητήρια στην κυρία Μακλάρκιν για, την, ε, για τις ιδέες της, για την ε, ευρεία προσέγγιση. Αν δούμε τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας των διαφόρων χωρών, βλέπουμε δυστυχώς διαφορετικά συστήματα με διαφορετικό υπόβαθρο, ιστορική εξέλιξη, διαφορετικούς προϋπολογισμούς που διαφέρουν μεταξύ κρατών μελών σημαντικά και υπάρχουν και διαφορετικοί κανόνες σε διάφορους τομείς. Σύμφωνα με τις συνθήκες όμως παράλληλα, η υγεία και η οργάνωση της υγείας είναι θέμα εθνικό. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν μπορούν να κάνουν και πολλά σε αυτό το θέμα. Παράλληλα όμως, Μπορούμε να σκεφτούμε κάποιες δράσεις για να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες στην υγεία. Μπορούμε να δημιουργήσουμε κοινέ στρατηγικές καταπολέμησης διαφόρων νόσων. Επίσης μπορούμε να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές μεταξύ κρατών μελών και μπορούμε να ενθαρρύνουμε από το ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Κομισιόν, να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν αυτές τις βέλτιστες πρακτικές. Όταν μιλάμε για την προστασία καταναλωτών, για παράδειγμα, κατά της ε, κακής ε, πρακτικής. Αυτό δεν είναι το ίδιο σε όλες τις χώρες μέλη δυστυχώς, οπότε και εδώ υπάρχουν ανισότητες. Είναι καθήκον μας λοιπόν να δημιουργήσουμε κάποια ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας καταναλωτών σε περίπτωση ε, κακής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Ε, επίσης ενημέρωση των ασθενών μπορεί να παίξει ρόλο κατά των ανισοτήτων. Και τέλος ε, η οδηγία για τη διοσυνοριακή ιατρική περίθαλψη, ε, φροντίδα για την υγεία, ώστε οι πολίτες ε, να επιδιώκουν την καλύτερη αγωγή. Και αυτό μειώνει τις ανισότητες. Και αύριο περιμένω θετική ψήφο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και μια συμφωνία με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπούσο για τους ε, πρασίνους. Ε, θα μιλήσω εγώ, είμαι σκιώδης, θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ την ε, εισηγήτρια για τις προτάσεις και τους σκιώδης για τις σημαντικές παρατηρήσεις. Είναι, ήταν πολύ καλή αυτή η σημερινή συζήτηση για το θέμα μας. Καταρχήν στηριζόμεθα σε θέματα που εντάσσονται σε αυτή την έκθεση γιατί η διασυνοριακή φροντίδα για την υγεία ρυθμίζεται κάπου αλλού. Οπότε δεν θα κάνουμε διπλή δουλειά, θα επικεντρωθούμε εμείς εδώ σε αυτά που μπορούμε να ρυθμίσουμε μέσω αυτής της έκθεσης. Τα βασικά είναι το θέμα ενημέρωση, πρόληψη. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν στην έκθεση αυτή. Αυτές τις σύντομες παρατηρήσεις είχα να κάνω ως σκιώδης και τώρα ως πρόεδρος, βάζω το καπέλο της πρόεδρου και δίνω το λόγο στον κύριο Ντε Ιζόγκ. Α, δεν θέλει να μιλήσει εξ ονόματος της Γκουε. Όχι. Ο κύριος Σαβίνη δεν είναι εδώ, οπότε περνάμε στα υπόλοιπα μέλη. Κυρία Σάλτεμπρος. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια για την εξαιρετική παρουσίαση. Συμφωνώ απολύτως ότι θα πρέπει να αγωνιστούμε περισσότερο, να κάνουμε περισσότερα πράγματα στον ε, τομέα αυτό. Ε, τουλάχιστον θα πρέπει να βελτιώσουμε την συλλογή και ανταλλαγή στοιχείων έτσι ώστε να ξέρουμε πού βρισκόμαστε στα διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχει και κάτι ουσιώδες ε, το οποίο δεν αναφέρθηκε όμως και που είναι ουσιώδης λέγω έτσι ώστε να έχουμε ε, ισοτιμία και ίσες συνθήκες ε, στην ε, τομέα, στον τομέα της υγείας. Αναφέρομαι στην κατάρτιση και την ενημέρωση. Όσο πιο καταρτισμένο θα είναι το ιατρικό προσωπικό, τόσο λιγότερες θα είναι οι ανισότητες στον τομέα της υγείας. Επομένως θα πρέπει να έχουμε μακροπρόθεσμες προοπτικές. Θα πρέπει να ε, ε, πείσουμε κιόλα τους νέους της Ευρώπης να ασχοληθούν με την κατάρτιση αυτή, να ασχοληθούν με τον ε, τομέα αυτόν και βεβαίως ε, ανταλλαγή πληροφοριών, ε, συλλογή στοιχείων, αλλά όλα αυτά να γίνουν μακροχρόνια έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο ε, όπου ο κάθε ένας πολίτης θα είναι καλά πληροφορημένος και ενημερωμένος. Η κυρία Στάιλερ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εισηγήτρια και τους σκιώδης. Νομίζω ότι η συνάδελφος που μίλησε προηγουμένως πραγματικά έθεσε το δάκτυλο από τον τύπο των ε, ύλων ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν ανισότητες στην τομέα της υγείας, όπως υπάρχουν και ανισότητες μεταξύ των ανθρώπων. Θα πρέπει με τον ίδιο τρόπο να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Και ε, βεβαίως αυτά που είπατε για την ε, ένδια, για τη φτώχεια, είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα είμαστε και στο ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και επομένως θα πρέπει να το προσέξουμε γι' αυτό. Ε, και θα πρέπει να γίνει έγκαιρα η παρέμβασή μας μίλησε ε, ο ε, σκιώδης ε, του ΕΛΚ για τις περικοπές που θα γίνουν και στο Ηνωμένο Βασίλειο στη δικιά μου χώρα θα γίνουν πολλές περικοπές και οι ανισότητες αντί να μειωθούν θα αυξηθούν. Μας ενδιαφέρει πολύ η προστιθέμενη αξία των συζητήσεων, των ανταλλαγών πρακτικών στην ε, Σκοτία ας πούμε εμείς έχουμε εισαγάγει την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος στην, στον, στο κάπνισμα ε, σε δημόσιους χώρους και μέσα σε τρία χρόνια, τέσσερα, έχουμε μείωση κατά 18% των περιστατικών αναπνευστικών προβλημάτων παιδιών ε, που φτάνουν στα νοσοκομεία. Και επομένως μας ενδιαφέρει η δημόσια υγεία πολύ, όχι μονάχα των παιδιών, η δημόσια υγεία γενικά. σχετικά με την πληροφόρηση, την ενημέρωση των ε, ασθενών. Πιστεύω ότι όντως θα πρέπει να ε, υπάρχει καλή ενημέρωση. Λίγο πριν είχαμε ε, συζήτηση σχετικά με την διαφήμιση και διαφήμιση φαρμακευτικών ε, προϊόντων. Ε, όταν αναφερόμαστε βεβαίως στην ενημέρωση των πολιτών, στην ενημέρωση των ασθενών, δεν αναφερόμαστε στην προπαγάνδα που θα κάνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να συζητήσουν και να αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα και προβλήματα τα σχετίζονται και με ειδικέ αρρώστιες. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε να συζητήσουμε όλοι μαζί και να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα. Μίλησε κάποιος για πρόληψη. Ίσως εσείς κυρία Πρόεδρε, ναι, ναι, ε, μιλήσαμε λοιπόν για πρόληψη, μα είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα η πρόληψη. Ας πούμε, ε, ασχολήθηκα πρόσφατα πολύ με τις ε, ε, αρρώστιες ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, των πνευμόνων, αυτές οι βροχίτιδες οι οποίες είναι πολύ συχνές, διαρκούν πολύ. Θα πρέπει να δούμε τι σημαίνουν, ας πούμε, οι βροχίτιδες αυτές για το σύστημα υγείας. Ε, και εάν είχαμε έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, δεν θα προχωρούσαν τόσο πολύ οι ασθένειες αυτές έτσι ώστε μετά να είναι δύσκολη και ακριβή η αντιμετώπιση τους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Στάιλερ. Η Κομισιόν, ο κύριος Πράις ζητεί το λόγο. Γιατί από τα άλλα παρόντα μέλη δεν ζητεί άλλο το λόγο. Κύριος Πράις, Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΙΜΚΟ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έδειξε ενδιαφέρον για την ανακοίνωση της Επιτροπής για τις Ανισότητες στον τομέα της υγείας. Εκτιμώ ιδιαίτερα τις παρατηρήσεις της εισηγήτριας αλλά και τις ε, παρεμβάσεις ε, των υπόλοιπων βουλευτών σήμερα. Μαζί με τον συνάδελφό μου από την ΓΔ για την απασχόληση είμαστε εδώ Κάτι που δείχνει ότι ήταν μια κοινή πρωτοβουλία των επιτρόπων που είναι αρμόδια για την υγεία και την κοινωνική πολιτική, που ήταν μάλλον στην προηγούμενη επιτροπή. Όπω είπαν και οι ομιλητέ, αυτό αντικατοπτρίζει την ανάγκη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε άλλες πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Όπως είπα, Υπάρχουν αχανείς ανισότητες, υπάρχει 14, 14 ε, ε, έτη διαφορά στο προσδόκιμο επίπεδο μεταξύ ανδρών και γυναικών, διαφορά 3 έως 5 ετών επίσης ό,τι αφορά το επίπεδο των επαγγελματικών ε, προσόντων που είναι ο μέσος όρος, φτάνει μέχρι και στα 10 χρόνια σε κάποια κράτη. Για τις ευάλωτες μάλιστα ομάδες σε αυτές οι διαφορές, παραδείγματος για τους Ρωμά, μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερες οι διαφορές. Η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λοιπόν που περιγράφεται στο έγγραφο είναι ότι τα αίτια, ναι, Πράγματι, ε, πολλά από αυτά τουλάχιστον μπορούν να αποφευχθούν. Καταρχήν, η σημαντικότερη ομάδα αιτίων βέβαια είναι κοινωνικο-οικονομικά. Πολιτικές για μεγαλύτερη τοπική εδαφική συνοχή, μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, μείωση της στόχιας από οικονομικής πλευράς, καταπολέμηση του αποκλεισμού. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι θεμελιώδη για την αντιμετώπιση του προβλήματος αλλά και οι σχετιζόμενες με την υγεία συμπεριφορές από τις οποίες ορισμένες ορθούνται από ε, οικονομικό μειονέκτημα όπως είναι η χρήση αλκοόλ ή το κάπνισμα παραδείγματος χάρη. Και βέβαια το σύστημα υγείας έχει το ρόλο του. Δεν τονίζεται όμως συγκεκριμένα ως βασικό καθήκον γιατί δεν είναι το σημαντικότερο αίτιο, δεν είναι η εξήγηση η βασική, έχει βέβαια το ρόλο, αλλά δεν είναι το βασικό. Σε ό,τι αφορά τώρα τις πολιτικές για την εσωτερική αγορά και την προστασία των καταναλωτών, είπατε ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη για την αντιμετώπιση των τομέα των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Το σημειώσαμε. Είπατε για την προστασία των καταναλωτών, γενικότερα για την υγειονομική περίθαλψη. Σημείωσα, παραδείγματο χάρη, ότι τα ατυχήματα είναι ο σημαντικότερος λόγος θανάτων μεταξύ των νέων. και διακίνηση κάποιων προϊόντων, δηλαδή κάποιε συμπεριφορέ που σχετίζονται με την υγεία έχουν να κάνουν και με τον τρόπο τη εμπορία και διανομή ορισμένων ε, προϊόντων. Η προστασία των ευάλωτων ομάδων, όπω προείπαμε, φυσικά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη. Βέβαια, μια εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά είναι πολύ σημαντική για την καταπολέμηση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας λόγω διαφορών ε, στην απόδοση των οικονομιών των κρατών μελών. Και βέβαια υπήρξαν πολλά ε, σχόλια για το σύστημα υγειονομικής περιθαλψής. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα αυτά. Ήταν σημαντικά αυτά που είπατε για τις τιμές των φαρμάκων, τις τιμές των ασθενών, στο τεφάλι καταγραφή των επαγγελματικών προσόντων, την μετακίνηση επαγγελματιών του κλάδου της υγείας. η ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κρατημέλη και όλε οι περιοχέ των κρατομελών να μπορούν να προσλαμβάνουν αλλά και να διατηρούν προσωπικό υψηλού επίπεδου. Ιδίως όταν ξέρουμε ότι διαφέρουν σημαντικά οι πόροι που είναι διαθέσιμοι. Φυσικά και επιθυμούμε να συνεργαστούμε με την Επιτροπή σας, αλλά και με τα κρατημέλη τα οποία είναι υπεύθυνα για την διαχείριση και την, ε, ε, των συστημάτων υγείας και την παράδοση αποτελεσμάτων. για να συνεχίσω. Θα δώσω το λόγο στον ε, συνάδελφό μου, αν δεν έχετε αντίρρηση, κυρία Πρόεδρε, ο οποίο θα σας μιλήσει και για τον ρόλο της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας για την προαγωγή, για την προώθηση της πρόσβασης στα συστήματα της υγειονομικής περίθλιψης και στη των ανισοτήτων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο για να συμπληρώσω αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος Just Price. Πράγματι, η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας συμμετέχει ενεργά στο ζήτημα αυτό. Βέβαια, η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας είναι ένας φορέας συνεργασίας πάνω απ' όλα, συνεργασίας μεταξύ του ευρωπαϊκού επίπεδου και των κρατών μελών. Γιατί μιλάμε για ένα τομέα που κατά προτεραιότητα βέβαια αφορά τα κράτη-μέλη. Πάντως, η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας στη γνωμοδότησή της στι 18 Μαΐου σημείωσε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τα διάφορα σημεία που αναφέρονται στην ανακοίνωση και συγκεκριμένα, όπως υπογραμμίστηκε και με τους, από τους διάφορους παρεμβαίνοντες, τη σημασία των ευάλωτων ομάδων, των ευαίσθητων ομάδων, γιατί πράγματι έχουμε να κάνουμε με ανισότητες στον τομέα της υγείας, αλλά και με γεωγραφικές ανισότητες, ανισότητες μεταξύ χωρών αλλά και εντός κρατών μελών και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Έχουμε όμως επίσης να κάνουμε και με ένα πιο ιδιαίτερο πρόβλημα, το οποίο αναφέρει και περιγράφει εντελεχώς και η επιστημονική έρευνα και αυτό που είπε η συγκίτρια για την έρευνα που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει να κάνει με τις ευάλωτες ομάδες. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην ε, περίθαλψη, εδώ και κάποια χρόνια, το 2006 συγκεκριμένα, η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Απασχόληση Κοινωνική Υποθέσεις συμμετέχει πιο ενεργά σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας και αυτό που εμείς λέμε οικονομική βιωσιμότητα των ε, συστημάτων υγειονομικής πέθαψη στο πλαίσιο της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού. Είμαι πεπισμένος για την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την κατεύθυνση αυτή. Συνάγοντας λοιπόν συμπεράσματα, η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας αποφάνθηκε υπέρ της υλοποίησης μέτρων με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης ε, στα συστήματα υγείας. Στις 18 Μαΐου λοιπόν εξέδωσε αυτή την επίσημη νομοδότηση. Η ανταλλαγή δεδομένων επίση, η ανταλλαγή πληροφοριών είναι πολύ σημαντική. Μεταξύ των διαφόρων δράσεων παρακολούθησης που αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπή, η ανταλλαγή δεδομένων και η βελτίωση τη συλλογή δεδομένων, εφόσον πρόκειται για την κοινωνική διάσταση, κοινωνικο-οικονομική διάσταση, είναι προτεραιότητα. Και δι ο καθορισμός δικτών δικτών που βέβαια θα πρέπει εν συνεχεία να επικυρωθούν από τις αρμόδιες αρχές. Αλλά τα τελευταίους μήνες πράγματι εργαστήκαμε πολύ και συνεργασία με την Eurostat και με τα κράτη-μέλη για την αρμοδιότητα των κρατών μελών. Συνεργαστήκαμε λοιπόν και επεξεργαστήκαμε ακριβώ αυτό το ζήτημα συλλογή δεδομένων κατάρτιση δικτών. Σε ό,τι είπε λοιπόν και ο Τσάστ Price, να προσθέσω ότι από στρατηγική σκοπιάς αυτό που είναι σημαντικό είναι η ενσωμάτωση της υγείας σε όλες τις πολιτικές. Δηλαδή όλες οι πολιτικές πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας του πολίτη. Γιατί νομίζω ότι πραγματικά δεν έχουμε να κάνουμε ένα κλινικό θα έλεγα πρόβλημα. Μακροπρόθεσμα λοιπόν όλοι οι καθοριστικοί παράγοντες από κοινωνικής πλευράς και όλη η πορεία ε, της ζωής κάποιου θα καθορίσει και το πώς θα εξελιχθεί η υγεία του. Ευχαριστώ. Η εισηγήτρια τώρα. Παρακαλώ, κυρία Μακλάρκιν, να ε, μας πείτε και για το χρονοδιάγραμμα που προτείνετε. Ευχαριστώ τους Σκιώδης και όλα τα μέλη και την Κομισιόν για τα σχόλια επί της εκθέσεως. Ευχαριστώ που είπατε ότι ήταν ευρεία η προοπτική που υιοθέτησα. Ήθελα να προσθέσω και άλλα θέματα, γιατί είναι κορυφαία η προτεραιότητα. Κέριος ο τομέας, υγεία, παιδεία, τα πιο σημαντικά. Όσο πιο πολύ το κοιτάζει κανείς, τόσο πιο πολύ ενδιαφέρεται και θέλει να συμπεριλάβει πράγματα. Εγώ ήθελα να δω βέβαια το, την πτυχή της εσωτερικής αγοράς ίσως είδα με περιοριστικό τρόπο τα αίτια της κατάστασης γιατί πάντοτε ήθελα να επικεντρώνομαι στην εσωτερική αγορά σε σχέση με την υγεία. Άκουσα πολλά ε, ε, σωστά πράγματα τα οποία θα συμπεριληφθούν όμως και στην έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος που θα επεκταθούν περισσότερο. Εμείς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες και τους οικονομικούς δείκτες ε, που διέπουν τις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Αυτά πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Τα ερευνητικά προγράμματα αναφέρθηκαν, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με την αγορά ώστε να φροντίσουμε ότι οι επενδύσεις θα συνεχιστούν. Γιατί είναι πολλές οι επενδύσεις και πρέπει να φροντίσουμε ότι θα εξακολουθήσει στην έρευνα και την ανάπτυξη να είναι κορυφαία. Ε, η ε, Ευρώπη στο μέλλον είναι όμως αρμοδιότητα κρατών μελών, θα πρέπει να δούμε τι έχουμε. Μπορεί να είναι ένα χωνευτήρι η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συλλογή αυτών των νέων ιδεών, των ε, βασικών κατευθυντηρίων και βέλτιστων πρακτικών. Όλα αναφέρθηκαν σήμερα το πρωί. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε πάλι την, ε, το ρόλο που μπορεί να παίξει η εσωτερική αγορά ως Επιτροπή για την εσωτερική αγορά το χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρω ακριβώς πότε λάβατε τις μεταφράσεις, αλλά 7-12 είναι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. 10 Νοεμβρίου θα υποβληθεί, οπότε σε μία εβδομάδα περίπου θα έχετε τις μεταφράσεις σας. Θα εξεταστεί 29 και 30 Νοεμβρίου η έκθεση, ή 30 7 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών και 10 Ιανουαρίου η ψηφοφορία. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Το λιανικό εμπόριο. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτη, η συγγήτρια, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα θυμάστε ότι στις 29 Σεπτεμβρίου στην τελευταία μας συνάντηση η Επιτροπή παρουσίασε μια πολύ καλή ανάλυση σχετικά με τον ελληνικό εμπόριο, χωροθετώντας τα προβλήματα τα οποία είχαν προκύψει στη συζήτηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Έγινε και η συζήτησή μας σχετικά με στέρνους ανταγωνισμού, έλλειψη διαφάνειας, ε, έλλειψη προσβασιμότητας των πελετών ε, στα κέντρα πώληση κτλ. Και μετά είπαμε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε σε κάποια ε, σημεία ε, ε, προτεραιότητας. Θα είναι τέσσερις σελίδες η έκθεση και δεν θα προσθεθεί τίποτα σε αυτό. <clears throat> Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε μια έκθεση η οποία θα είναι προσανατολισμένη προς συγκεκριμένε δράσεις και που θα αντιμετωπίζουν τα κύρια προβλήματα τα οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη κατέδειξαν. Συγκεκριμένα παραδείγματα, ε, συγκεκριμένε περιπτώσεις ακόμα, έτσι ώστε να μας ε, οδηγήσει σε καλύτερη λειτουργία στο λιανικό εμπόριο. Πρώτη φορά ασχολούμαστε με τέτοιο συνολικό τρόπο στο λιανικό εμπόριο. Ε, είναι ένα εμπόριο όμως το οποίο συμμετέχει συμμετέχει στην ανάπτυξη της Ευρώπης, δημιουργεί θέσει εργασία και επομένως είναι κάτι σημαντικό. Στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συνάντηση με τους κοιόδη ηγητέ και τους ευχαριστώ εν παρόδο για την επικοδομητική τους ε, συνέργεια. Επίσης, ε, ε, είχα εκφράσει την επιθυμία για ευρύτερη διαβούλευση, γι' αυτό ήθελα και περισσότερο χρόνο. Ε, τώρα, ποιες ε, είναι η καταπροτεραιότητα, ποιοι είναι η καταπροτεραιότητα τομείς. Καλύτερη προσβασιμότητα στα μαγαζιά ε, και στα προϊόντα, στα αγαθά από των καταναλωτών η άρση των περιορισμών. Υπάρχουν ακόμα πολλοί περιορισμοί ε, στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών. Όσο τρελό και αν ακούγεται, ακόμα υπάρχουν. Ε, ας πούμε κάποια κρασιά τα οποία θέλουν συγκεκριμένο πιστοποιητικό τυριά που δεν μπορούν να εξαχθούν παρά μόνο εάν υπάρχουν ε, συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Νομίζω ότι εμείς εδώ δεν θα ε, επανανακαλύψουμε τον τροχό, αλλά μέσω ανταλλαγής απόψεων θα μπορέσουμε ε, να ε, δούμε ποια είναι τα προβλήματα και ενδεχομένως να αρθούν κάποιοι περιορισμοί της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και βεβαίως θα μπορέσουμε ενδεχομένως να ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να συνεργαστούν μαζί μας. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο προέκυψε είναι οι περιοριστικές πρακτικές ε, οι οποίες περιορίζουν ε, την επιλογή και κρατούν τις τιμές ψηλά. Σε πολλούς τομείς σε πολλούς ε, για να μπορέσουν να προωθήσουν κάποια προϊόντα στο λιανικό εμπόριο δίνονται κάποιες, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, κάποιοι περιοριστικοί όροι. Τέλος, ε, ένα άλλο ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό είναι η επίπτωση στο περιβάλλον, οι συσκευασίες και η επίπτωση που έχουν στο περιβάλλον. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να δούμε την καινοτομία. Υπάρχουν ε, επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εξαιρετικά μεγάλες δυνατότητες για έρευνα και ε, ανάπτυξη και νομίζω ότι θα είναι προς όφελος όλων εάν χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη αυτών των επιχειρήσεων. Ε, βεβαίως ε, θέλουμε οι αποφάσεις να παίρνονται σε κοινοτικό επίπεδο και αναφερόμαστε εδώ σε ζητήματα τα οποία αφορούν το κοινοτικό επίπεδο και όχι το τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Μεγάλο μέρος της δουλειάς μας δεν είναι να προτείνουμε ε, κανονισμούς ή νομοθεσία αλλά ίσως να προτείνουμε ακριβώς ότι δεν χρειάζεται κανονιστική ρύθμιση για ένα συγκεκριμένο ε, περιβάλλον. Και έρχομαι σε κάτι που όλοι αναφέρουν. Ε, μη ε, σωστές εμπορικές πρακτικές. Αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός, χρήση αθέμητων πρακτικών, είναι κάτι που ενδιαφέρει όλους. Νομίζω ότι θα πρέπει στην ε, συζήτηση να ε, βάλουμε θέματα τα οποία μέχρι τώρα ο κόσμος φοβάται να τα αναφέρει. Χρειαζόμαστε διάλογο, χρειαζόμαστε εταιρική σχέση με τη βιομηχανία. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτήν την πρακτική κατηγόρου ενδεχομένως που είπαμε μέχρι τώρα και που πολύ συχνά ε, μπλοκάρει τελικά την ε, δυνατότητα διαλόγου και επομένως εξέβρεσης επικοδομητικών λύσεων. Ε, υπάρχει και θα πρέπει να αφήσουμε χώρο για την αυτορύθμιση, για την εθελοντική ρύθμιση. Και τελικά η έκβαση ο ρόλος που θα παίξει αυτή η έκθεση είναι να, μας, να δούμε πόσο, κατά πόσον ε, η βιομηχανία θέλει να πάρει εθελοντικές ε, ε, δράσεις, θέλει να αναλάβει εθελοντικά κάποια μέτρα, πόσο θέλει να συζητήσει και να έχει διάλογο μαζί μας. Χρονοδιάγραμμα. Ζήτησα από τη Γραμματεία λίγο περισσότερο χρόνο γιατί νομίζω ότι σημαντικό για το αποτέλεσμα είναι να ενσωματωθούν στην διαδικασία αυτή όσο γίνεται περισσότεροι. Μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις, ε, κοινωνία των πολιτών, ε, εκπρόσωποι. Στις 30 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει τη δικιά της ε, διαβούλευση. Συγγνώμη, 27 Οκτωβρίου λέει η ομιλήτρια, θα κάνει την δικιά της διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη Ανοιχτέ οι πόρτε για όλους και στις 3 ε, ε, Νοεμβρίου θα, κάνουμε, θα οργανώσουμε ένα εργαστήριο, ένα workshop. Ε, δεν έχουμε ακόμα κατασταλάξει πώς θα είναι, ποια θα είναι η μορφή. Θα κάνουμε μια συζήτηση στη Σουηδία, είναι ευρωπαϊκή συζήτηση και όλοι είναι καλοδεχούμενοι. Συμφώνησα με την Γραμματεία να υποβάλω την παρουσία στην έκθεσή μου αρχές Μαρτίου ε, και να ε, προχωρήσουμε σε ψηφοφορία στα μέσα Απριλίου όταν θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία. Έχω έρθει ήδη σε επαφή, έχω συζητήσει το θέμα με του σκιώδη αλλά βεβαίως περιμένω και τα σχόλιά σα όσον αφορά και το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία. Ο κύριος Χάμπερ με εξουσιοδότησε να πω κάτι για το χρονοδιάγραμμα, ότι το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ γενναιόδωρο πάει πολύ μακριά και θα έχουμε πρόβλημα να συντονίσουμε και άλλα θέματα όπως το πακέτο για την εσωτερική αγορά. Καλό είναι να το κάνουμε λίγο πιο σφιχτό το χρονοδιάγραμμα. Ο Σχιώδης το κατανοώ ότι χρειάζεται μακρότερος χρόνος διαβουλεύσεων, αλλά ως πρόεδρος, γιατί φοράω δύο καπέλα, διαπιστώνω ότι ενδεχομένως θα έχουμε προβλήματα με τις άλλες μας δουλειές. Θα το συζητήσουμε αυτό επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Γκέπ Χάρτ που εκπροσωπεί τον κύριο Πανσέρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Κοράτσα Μπίλτε για τις εξε... εκτενείς παρατηρήσεις Ο κύριος Παντσέρη θεώρησε την συνάντηση της περασμένης εβδομάδας πολύ επικοδομητική και ευχαριστώ και εξ ονόματός του. Για το χρονοδιάγραμμα τώρα. Συμφωνώ με το σχόλιο που μετέφερε η πρόεδρος από τον κύριο Χάρμπορ. Εμείς ως συντονιστές στο ΙΜΚΟ αποφασίσαμε στο πακέτο για την εσωτερική αγορά να καταρτήσουμε τρεις εκθέσεις που θα τρέξουν παράλληλα και δεν θα διαχωριστούν. Αλλά για κάτι τέτοιο χρειάζεται να έχουμε τις ελεύθερες ε, θέσεις που θα ελευθερωθούν και από το γεγονός ότι θα τελειώνουν γρήγορα οι εκθέσεις. Οπότε πρέπει πραγματικά να ξανασυζητήσουμε το χρονοδιάγραμμα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εδώ ώστε να τα προλάβουμε όλα όσα αποφασίσαμε. Επί της ουσίας. Συμφωνώ σχεδόν με όλα. Με όλα ουσιαστικά γιατί αναδείξατε και καταδείξατε τα προβλήματα πολύ καλά, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ότι θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα ώστε οι μικρές επιχειρήσεις να έχουν και αυτές μια ευκαιρία να ζήσουν και να επιβιώσουν στο σημερινό αυτό είναι πολύ μεγάλη φροντίδα δικιά μας. Όχι μόνος γιατί θεωρούμε ότι τα καταστήματα αυτά από μόνα τους είναι σημαντικά, αλλά επειδή έχουν μεγάλη σημασία και για τους καταναλωτές. Και θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε ώστε οι υπηρεσίες ε, που προσφέρουν συνίστανται στο ότι είναι κοντά τα καταστήματα αυτά στον κόσμο για τις αγορές. και φροντίζουν στο να μπορεί, μπορούν να ασκούν την αγοραστική τους δυνατότητα οι καταναλωτές. Σημαντικό είναι επίσης το θέμα της αστιφιλίας και οι κανόνες που θεσπίζουμε για να διασφαλίσουμε ε, ότι δεν θα υπάρχει υπερβολικά μεγάλος, βλέπε αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων και μικρών. Θα πρέπει δηλαδή να διατηρήσουμε τις ευκαιρίες των μικρών. Και ένα άλλο θέμα το οποίο θίξατε είναι η πρόσβαση στην αγορά. Πράγματι, Πρέπει να το καταπιαστούμε αυτό το θέμα, όπως, και, όπως κάναμε και με την οδηγία για τις υπηρεσίες. Πρώτα χρειάζεται ε, μια πρώτη εξέταση του θέματος, ένα screening. Τι λογική, ποιοι λογικοί κανόνες υπάρχουν, γιατί υπάρχουν και λογικοί και σωστοί κανόνες, υπάρχουν και άλλοι όμως που μας κάνουν να αναρωτιόμαστε τι σχέση έχουν αυτοί με την ποιότητα του εμπορίου. Ε, έχουμε και προστατευτικά μέτρα θέλω να πω και πρέπει να τα καταπολεμήσουμε γιατί εμείς θέλουμε μια γνήσια εσωτερική αγορά στον τομέα αυτό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι ε, θίγεται το ζήτημα αυτό. Για μας τους σοσιαλδημοκράτες το άνοιγμα της αγοράς δεν σημαίνει ε, αναρχία και απορρίθμιση, η κατάργηση όλων των ρυθμίσεων, αλλά συνετή και σωστή ρύθμιση. Όχι το λέω αυτό για να μην παρεξηγηθούμε σε ό,τι αφορά αυτά τα δύο θέματα. Επίσης, σε αυτά τα πλαίσια πολύ θα πρέπει να μας απασχολήσει και κάτι ακόμα. Ότι δηλαδή το λιανικό εμπόριο θα πρέπει να λειτουργεί και σε μικρές περιοχές για, γιατί έχει σημασία ε, για ιδιαίτερε κατηγορίε του πληθυσμού, ηλικιωμένοι, άνθρωποι περιορισμένη, κινητικότητα, ε, ακόμα και όταν πρόκειται για διαδικτυακέ αγορέ, δεν αποτελεί αυτό λύση για όλους. Σκέφτομαι για παράδειγμα ότι οι ηλικιωμένοι κυρίως, ε, υπάρχουν ηλικιωμένες γυναίκες που ζουν μόνες, οπότε εκεί Υπάρχει και ένα θέμα κοινωνικό, ψυχολογικό, ότι δεν μπορεί δηλαδή να αναγκάζονται μόνο να αγοράζουν από το διαδίκτυο, αλλά να έχουν και μια κοινωνική ένταξη βγαίνοντα για να κάνουν τις αγορές τους σε κάποιο κατάστημα και αυτό πρέπει να το δούμε. Οπότε πρέπει επίσης πολύ συγκεκριμένα να σκεφτούμε πώς μπορούμε ουσιαστικά να προσφέρουμε βοήθεια στις επιχειρήσεις αυτές. Τα μπέρδεψα τώρα, Πιτέλα ε, Παντσέρη, όχι, ο κύριος Παντσέρι, είναι, ο κύριος Παντσέρι. Ε, προτείνει να σκεφτούμε ίσως και φορολογικά μέτρα για να ε, τους ελαφρύνουμε. Και αυτό είναι κάτι που αξίζει να συζητηθεί και να εξεταστεί, ώστε να είναι ανταγωνιστικές αυτές οι επιχειρήσεις. Και κάτι ακόμα επίσης, που δεν μου το πω ο κύριος αλλά που εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις η διαφάνεια των ενοικίων που ζητούνται. Πολλές φορές τα ενίκια είναι εξωφρενικά που τσακίζουν τις μικρές κυρίως επιχειρήσεις. Και γι' αυτό ε, θα πρέπει να το δούμε, γιατί μετά κλείνουν. Ε, υπάρχει λοιπόν και μια έντονη παράμετρος εδώ της γενικότερης πρόνοιας που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Πρόκειται για υπηρεσίες, προσφορές γενικού ενδιαφέροντος που έτσι θα πρέπει να ειδωθούν πολλές από αυτές τις ε, ε, υπηρεσίες αυτών των καταστημάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούκεγκάρτ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ο κύριος Λούκεγκάρτ ε, συνοδεύεται από τη Δανέζικη τηλεόραση. Ε, έχετε το, λόγο, δεν νομίζω να έχουμε κανένα πρόβλημα. Έχετε όλη την κατανόηση. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη γιατί ήρθα λίγο αργοπορημένος και έχασα το πρώτο μισό της παρέμβασης της κυρίας ε, ε, Μπίλτ. Ενδεχομένως λοιπόν από πράγματα που τα έχουμε ήδη πει. Ε, πρώτα απ' όλα έχουμε ένα έγγραφο το οποίο μας έχει υποβληθεί και στην ουσία δεν αναφέρονται εκεί οι προτεραιότητες που είχαν απορρεύσει από την συνάντηση της, με την Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σαφές για μας ότι θα πρέπει να έχουμε προτεραιότητες και να αναφέρονται αυτές. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να περιοριστούμε ε, σε θέματα τα οποία αφορούν την εντολή της Επιτροπής ΙΜΚΟ. Δεν νομίζω ότι ε, πρέπει να ξεπεράσουμε ε, την εντολή της Επιτροπής αθέμητες πρακτικές ε, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει πριν ε, συμφωνήσουμε για οποιουσδήποτε κανόνες ε, θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη έρευνα αντικτύπου γιατί ξέρετε μπορεί να τελικά να οδηγηθούμε σε προβλήματα όσον αφορά την λυσίδα διανομής. Δεύτερον, θέλουμε μια εσωτερική αγορά η οποία να λειτουργεί καλά. Ε, αυτή τη στιγμή ε, μιλάμε για γεωγραφικούς περιορισμούς προμήθειας. Ε, πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Θα πρέπει να δούμε τις διαφορές που υπάρχουν στις τιμές ε, για τα ίδια προϊόντα ανάμεσα σε κράτη-μέλη γιατί ενδεχομένως κάποιοι επιπλέον δασμοί, ψηλός ΦΠΑ μπορεί να προκαλεί τις ε, αλλαγές αυτές και επομένως ε, θα πρέπει να το δούμε. Επίσης ε, να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο. Φυσικά θα πρέπει να δούμε ε, όλο το σύστημα αυτό στα πλαίσια ε, της ε, νέας όθησης που θέλουμε να δώσουμε στην, ευρωπαϊκή, στην εσωτερική αγορά. Επίσης, ανταγωνισμός όσο και, όσο όλο και περισσότερες είναι οι ιδιωτικές ετικέδες οι ε, ιδιωτικές ετικέτες οι οποίες περιορίζουν όλο και περισσότερο το χώρο που έχουν ε, οι άλλοι παραγωγοί γιατί βεβαίως οι μεγάλες φίρμες έχουν μεγάλη ευκολία στο να έχουν την δικιά τους ε, ιδιωτική ετικέτα. Αυτό όμως στενεύει, τον περιορίζει τον ανταγωνισμό. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν κάποια στοιχεία του εθνικού νόμου οποίο θα πρέπει, ε, τα, ε, τα οποία θα πρέπει να διατηρήσουμε. Αυτά είναι τα σημεία που ήθελα να θίξω και βεβαίω χαίρομαι που έχουμε στενή συνεργασία με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εγώ είμαι σκιώδης των Πρασίνων. Ευχαριστώ την εισηγήτρια θερμά για τη δουλειά μέχρι τώρα και για τη συνεργασία και για τη συνάντηση στο Στρασβούργο που βοήθησε νομίζω πολύ. Εμένα με ενδιαφέρει κυρίως εδώ να δούμε μήπως χρειαζόμαστε για το B2B, για τον τομέα Β2Β, για αυτό το τομέα, για τον αθέμητο ανταγωνισμό. Θα πρέπει να το δούμε, να μαζέψουμε στοιχεία αλλά είχαμε συζητήσει στα πλαίσια της ε, οδηγίας των ανταγωνισμού που έπρεπε να συμπεριλάβουμε τον τομέα Β2Β. Υπήρχαν πολλοί λόγοι. Η Κομισιόν αποφάσισε όχι, δεν ήθελε να το συμπεριλάβει τότε, αλλά νομίζω ότι η συζήτηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Και ένας στόχος ε, αυτής της έκθεσης είναι να ξαναδούμε τα προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα σε πολλούς τομείς που αυξάνονται, γιατί οι αλυσίδες μεγαλώνουν όλο και περισσότερο και δεν μπορεί το λιανεμπόριο να τη συναγωνιστεί επίσης ώρες ιδιαίτερα ε, στον ε, καινοτόμο τομέα, στις καινοτομίες εκεί παίζει μεγάλο ρόλο αυτό η διαφορά λιανεμπορίου μεγάλων αλυσίδων εφοδιασμού να δούμε λοιπόν αυτό το θέμα να δούμε όλες τις αθέμητες πρακτικές, να τις καταγράψουμε και να αρχίσουμε μια συζήτηση για το τι ρύθμιση ενδεχομένω χρειάζεται. Ως πρόεδρος πάλι ο κύριος De ο οποίο εκπροσωπεί τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν μπορεί να είναι παρόν ο συνάδελφος. Θα ζητούσα βέβαια ούτως ή άλλως το λόγο, γιατί πραγματικά χαίρομαι που η Επιτροπή συνέταξε την έκθεση αυτή σε μια επιστολή προς τον Επίτροπο Μπαρνιέ του είχα πει ότι η πρωτοβουλία αυτή ήταν πάρα πολύ καλή. Επίσης είχα αναφέρει στην επιστολή μου κάποια στοιχεία ε, σαν αυτά τα οποία μας ε, παρουσίασε η κυρία Γκέμπχαρτ. Το κοινωνικό λειτουργήμα των μικρών καταστημάτων αναφέρεται και είναι και πολύ σημαντικό και για μας. Αν δει κανείς την κατάσταση και τις εξελίξεις Βλέπουμε ότι τα καταστήματα μετακινούνται προς τα έξω, στα περίχωρα των πόλεων. Ε, η τοπική κοινότητα πολλές φορές ε, δεν είναι σύμφωνη και έχουμε και κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά κοινωνικές αξίες αλλά και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Η διάσταση της ασφάλειας είναι σημαντική και νομίζω ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί η σημασία της. Και εδώ έρχομαι να συμφωνήσω και με άλλους από τους προλαλήσαντες, ότι δηλαδή ε, είναι σημαντικό να υπάρχει αυτό το μαγαζάκι της γωνιάς, ε, το μαγαζάκι του χωριού. Πρέπει να το υποστηρίξουμε. Αυτή τη στιγμή λίγο πολύ κανείς είναι υποχρεωμένος να εργάζεται σε μια λυσίδα λόγω της οργάνωσης ε, των αγορών. Πρέπει να είναι κάποιος μέλος μιας μεγάλης αλυσίδας. Και αυτό που πολύ συχνά συμβαίνει είναι ότι πηγαίνει ο κόσμος σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ με το αυτοκίνητό του, γιατί αυτό, μάλιστα και αυτό δεν είναι καλό για το περιβάλλον, γιατί είναι πολύ πιο ακριβό το τοπικό ε, κατάστημα το μαγαζί της γειτονιάς. Και γι' αυτό και οι αυτοαπασχολούμενοι, οι λιανοπολιτές δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Υπάρχουν και κάποιες αθέμητες εμπορικές ε, πρακτικές, όπως είπατε, και αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και στο το business to business. Πιστεύω ότι κάποιες διευκολύνσεις θα πρέπει να δίδονται στα μικρά καταστήματα για να μπορέσουν να παραμείνουν, να διατηρηθούν στην Ήπεθρο. Δεν ξέρω αν θα, μπορούσαμε να τους παραχωρη... να... θα μπορούσαν να τους παραχωρηθούν κάποιες πιστοτικές διευκολύνσεις ε, ή κάτι ανάλογο. Δεν ξέρω, μήπω θα έπρεπε επίση να εκπονηθεί μια ξεχωριστή έκθεση, ένα σχέδιο δράση από την Κομισιόν για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να βοηθηθούν τα μικρά καταστήματα. Ο Επίτροπος όταν τον ρώτησα μου είπε ότι παρακολουθεί πολύ στενά τη συζήτηση που έχουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Ίσως λοιπόν στα μικρά αυτά ε, μαγαζιά, στα χωριά ή στις γειτονιές θα μπορούσαμε να τους δώσουμε ένα πιο ενισχυμένο ρόλο. Αυτό θα ήταν θετικό. Κύριος Ροσφόρ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Με τον Φιλίπ Σιβέν πριν μιλούσαμε για το αλκοόλ. Δεν θα πρέπει να πέσουμε στην παγίδα και για αυτό το θέμα ε, στον αλκοολικό που ψάχνει το βράδυ τα κλειδιά του μέσω σκοτάδι και ενώ είναι στο πρεβάζι αυτός το ψάχνει κάπου αλλού. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τη συζήτηση αυτή που έχουμε γιατί νομίζω δείχνει πάρα πολύ καλά ότι θέλουμε τελικά να διευρύνουμε το πεδίο. Δηλαδή πρέπει να έχουμε και προτεραιότητες αλλά ούτε και να παγιδευτούμε σε μια συζήτηση η οποία ουσιαστικά περιορίζεται στην συλλογή στοιχείων ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια των καταναλωτών. Κάτι που είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι και το παν. Στην εισαγωγή αυτού του consumer ε, scoreboard ε, λέγεται ότι οι καταναλωτές στην αρχή λέγεται ότι η ικανοποίηση των καταναλωτών πρέπει να είναι στο επίκεντρο των μελλοντικών ε, μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο εσωτερική αγορά. Σε όλε τι συζητήσει που είχαμε και τι οποίε θεωρώ πάρα πολύ σημαντικέ και για τον ανταγωνισμό και για τα μικρά καταστήματα, όπως έχει το scoreboard, ε, δεν απορρέουν κάποια θετικά στοιχεία, ούτε και ο καταναλωτής εκτιμά θετικά κάποια πράγματα. Παραδείγματος χάρη ό,τι αφορά ε, τον ανταγωνισμό. Πολύ συχνά ο καταναλωτής δεν γνωρίζει ότι κάποιε μεγάλε αλυσίδε που θεωρεί ανταγωνιστικέ θεσμένε προ τι ΔΕ, ουσιαστικά είναι θηγατρικέ του ίδιου ομίλου Και δεν κάνουν πραγματικό ανταγωνισμό μεταξύ του. Και ίσω ένα από τα πιο στρεβλά πράγματα που βλέπουμε σήμερα είναι αυτό. Σούπερ μάρκετ που είναι σε κοντινή απόσταση το ένα από το άλλο, αλλά φαίνεται να είναι σε διαφορετικέ αλυσίδε, αλλά είναι στον ίδιο όμιλο τελικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Επίσης θα πρέπει σε ό,τι αφορά τώρα την προστασία των μικρών καταστημάτων, πολύ ε, με ευχαρίστησε αυτό που είπαν οι συνάδελφοι, να ε, περασπιστούμε αυτά τα μικρά καταστήματα τη γειτονιά. Και εγώ είμαι υπέρ, αλλά πολλέ φορέ δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό, γιατί πολλές φορές θεωρούμε ότι δεν συνάδει η προστασία των μικρών καταστημάτων με την ε, ε, τήρηση των όρων του ανταγωνισμού. Νομίζω ότι θα πρέπει και μπορούν αυτά τα δύο να συνδεθούν μεταξύ τους και μακάρι να έχουμε συνένεση μεταξύ μας και να πούμε ότι θέλουμε να συνδέσουμε αυτά τα δύο μεταξύ τους. Έχω την εξή πεποίθηση, πολύ ισχυρή πεποίθηση, ότι πέραν της συσκευασία του τυριού και κάποιων άλλων αντιστοίχων θεμάτων, είμαι πεπισμένος ότι τα ζητήματα για τα οποία η ενημέρωση του καταναλωτή δεν είναι επαρκής, ότι ο καταναλωτής νομίζω ότι δεν είναι σαφή τα πράγματα στο κράτος με το οποίο μένει, νομίζω ότι είναι περίπου το ίδιο με κράτη τα οποία δεν διέπονται από καθεστώ εσωτερική αγορά. Να σα πω ένα παράδειγμα. Κινητή τηλεφωνία, τραπεζικέ υπηρεσίε. Πρόκειται για δύο τομεί που οι καταναλωτέ ε, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά του, ιδίω ό,τι αφορά το σύστημα τιμών. Και δεν είναι τυχαίο που για τα ίδια θέματα οι καταναλωτές έχουν την εντύπωση ότι είναι χειρότερα τα πράγματα όταν ε, χρειάζονται διασυνοριακές υπηρεσίες, τραπεζική υπηρεσία εκτός της χώρας στην οποία διαμένουν ή όταν πρέπει να χρησιμοποιήσουν το κινητό τους τηλέφωνο εκτός της χώρας στην οποία ζουν. Με άλλα λόγια, κάθε διευκρίνηση και διασαφήνιση του συστήματος τιμών εντός του κράτους μέλους συμβαδίζει με τη βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς χέρι-χέρι πάνω αυτά τα δύο. Αν υπάρχει αοριστία και αβεβαιότητα σε μία χώρα μέλος, αυτό επιδεινώνεται. Στην περίπτωση μετά που κάποιος θέλει να έχει ανταλλαγές που δεν θα πρέπει να υπονομεύονται και να υποσκάπτονται σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς. Και τώρα έχω ένα ερώτημα προς τον Ισίτη και τους, και τους Σκιώδης. Μας προτείνεται να δούμε ότι στα προσεχή στάδια για τη βελτίωση αυτού του πίνακα επιδός του scoreboard υπάρχει εντοπισμός 50 αγορών και λέω ότι δεν επαρκεί ο προϋπολογισμός για να παρακολουθούμε μαζί ε, συγχρόνως αυτούς τους 50 αγορές. μπορούμε να πούμε ότι θα παρακολουθούμε τις σημαντικότερες αγορές κάθε χρόνο και διαδοχικά ανάλογα με, τα, με το έτος θα βλέπουμε ε, τις επόμενες. Εγώ αυτό το οποίο θα προτιμούσα να έχουμε ένα σημείο για τις 50 αγορές, κάθε χρόνο όμως να επικεντρωνόμαστε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, να μην είμαστε διεξοδικοί κάθε χρόνο. Αυτό το προτιμώ να πούμε ότι δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε εξαντλητικά και πλήρω και διεξοδικά όλε τι αγορέ. Κάποιε από αυτέ τι τι παρακολουθούμε με κάποιου βασικού στρατηγικού δείκτε. Προτιμώ αυτό παρά να πούμε ότι παρακολουθούμε πλήρω και διεξοδικά τι αγορέ, αλλά όχι κάθε χρόνο. Γιατί υπάρχουν αγορέ, μίλησα για την κινητή τηλεφωνία, μπορώ να μιλήσω για το triple play και για τις τραπεζικές υπηρεσίες όπου λόγω της δυσκολίας να έχουμε πάρα πολύ πρόσφατα στοιχεία και χαίρομαι που ξαναείπαμε εδώ ότι θα ε, δοθεί ενθάρρυνση ε, να δουλέψει η Eurostat με τις στατιστικές των κρατών μελών κτλ. Αλλά δεδομένου του χρόνου που χρειάζεται για να συλλέξουμε τα δεδομένα και επειδή έχουμε κάποιε αγορέ που λέμε ότι δεν φιλοδοξούμε να τι παρακολουθούμε κάθε χρόνο, τελικά δεν θα έχουμε σχέση. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προτιμώ να πούμε και να έχουμε τον εξή στόχο. Εάν δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε δεξιωτικά όλε τι αγορέ κάθε χρόνο, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να παρακολουθούμε κάποια συγκεκριμένα στρατηγικά δεδομένα. Ευχαριστώ κύριε Ροσφόρη. Οι παρατηρήσει σα είναι σωστέ για το scoreboard και θα τι σημειώσουμε κατά τι εργασίε στο scoreboard αυτό το πίνακα βαθμολογία. Αλλά ε, εμείς αναφερθήκαμε προηγουμένως για την, στην ανακοίνωση της Κομισιόν για το λιανεμπόριο και θα μας πει σχετικά η Κομισιόν, αλλά οι προτάσεις να μην επανεφεύρουμε τον τροχό κάθε χρόνο για το σκόρμπορτ είναι πολύτιμη. Η κυρία Βερνιό είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την Αναμαρία. Μαρία και να κάνω μια μικρή παρατήρηση, μια σύντομη παρατήρηση που θα συνδέσει ε, την προηγούμενη συζήτηση για τη μείωση των ενισοτήτων στον τομέα τη Υγεία με το λιανικό εμπόριο. Η Επιτροπή ασχολήθηκε με ε, την ε, ανισότητα εγκατάστασης φαρμακείων στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κάθε πολίτης Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ίση πρόσβαση όχι μονάχα στην περίθαλψη αλλά και στα φάρμακα Μιλήσαμε για το εμπόριο στις, ε, στα μικρά χωριά, στις μικρές πόλεις ε, ε, και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ισόρροπη παρουσία των φαρμακείων και των μικρών φαρμακείων σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια και όχι να έχουμε φαρμακεία μονάχα στις μεγάλες πόλεις. Βλέπουμε ότι έχουμε παραπάνω φαρμακεία από όσα χρειαζόμαστε στις μεγάλες πόλεις και καθόλου στα χωριά ή στις μικρές πόλεις Πρόκειται για ένα θέμα δημόσιας υγείας, ασφάλειας των, ε, των ασθενών και επομένως ε, θα πρέπει τα φάρμακα να μπορούν, ε, αν δεν υπάρχει φαρμακείο, να μπορούν να διανέμονται ε, σωστά και όχι από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να δώσουν κάποιες συμβουλές υγείας στους ασθενείς. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σβάπε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακούμε, ακούσαμε πολλές διαφορετικές απόψεις. Είχαμε και μια γραπτή δήλωση της προηγούμενης ε, θητείας που έλεγε ότι οι μεγάλες ε, φύρμες ε, πολλές φορές στρεβρώνουν τον ανταγωνισμό χρησιμοποιώντας τη δύναμή τους με αθέμητο τρόπο. Είναι, είναι σίγουρα λοιπόν απαραίτητο να φτάσουμε σε μια σαφή θέση. Βεβαίως, βεβαίως ακούσαμε πολλά σχόλια ε, προς αυτή την κατεύθυνση ε, αλλά εγώ θα ήθελα να έχουμε μια πολύ σαφή ε, και δυνατή πάγια θέση πάνω στο θέμα αυτό όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα Ε, δεν μας ε, βοηθάει το χρονοδιάγραμμα, αυτό θα μας πάει στον επόμενο χρόνο. Δεν είναι δυνατόν και είμαι σίγουρος ότι η σχέδιες και η κυρία Μπίλτ θα βρούνε μια λύση όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Επίσης ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να... να δούμε και άλλα θέματα που συζητάμε τώρα, τον, τις ε, αθέμητες εμπορικές ε, πρακτικές ε, ανάμεσα στις επιχειρήσεις business to business, εμπορικές συναλλαγές business to business, όλα τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τους τηλεφωνικούς καταλόγους κτλ. Όσον αφορά το λιανικό εμπόριο θα ήθελα επίσης να πω το εξής. Κατά την άποψή μου, οι λιανέμποροι θα πρέπει ε, να ανεβούν λίγο στα μάτια του κόσμου. Ε, το εμπόριο είναι εμπόριο, είτε είναι μικρό, μεγάλο, λιανικό, χονδρικό ε, αλλά βλέπουμε ότι όλο και χάνεται το λιανικό εμπόριο. Οι μικροί έμποροι, οι λιανέμποροι σιγά σιγά εξαφανίζονται, κλείνουν. Δεν μπορούμε μόνο να ακολουθούμε τους ε, κανόνες της αγοράς, πρέπει μερικές φορές να τους δημιουργούμε κιόλας. Ε, ε, η κύριε Βηγό το είπε και θέλω να το αναφέρω κι εγώ. Η πρόσβαση των πολιτών στις, στα φάρμακα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν αφορά μονάχα θέματα αγορών, αφορά κυρίως θέμα δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας θα πρέπει να γίνουν σεβαστές κάποιες γενικές αρχές. η πώληση ολισμένων προϊόντων, η πώληση σε συγκεκριμένες τιμές. Είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Ε, θα ήθελα λοιπόν να διευρύνουμε όσο γίνεται το θέμα αυτό και για τα υπόλοιπα. Είμαι βέβαιος ότι η συγγήτρια και οι σκιώδης συγγήτρες θα κάνουν πολύ σωστές προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά και ακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον τη συζήτηση. Και παρακολουθούμε την εξέλιξη με την ένταξη τη έκθεσης. Αύριο ε, θα έχουμε μια, ε, ένα συνέδριο, μια συνδιάσκεψη μετά την έκθεση του Ελληνικού εμπορίου. 200 περίπου εμπλεκόμενοι θα είναι παρόντες και ελπίζω να συμπεριληφθούν τα αποτελέσματα της διάσκεψης αυτής και στα συμπεράσματα τη δική σας επιτροπή και θα συνεργαστούμε στενά μαζί σας γι' αυτό. Κάτι άλλο που θέλω να πω, και εδώ μιλάω με ειλικρίνεια, κυρία Πρόεδρε, εξακολουθώ να μην ξέρω τι θα έχει η πράξη της ενίας για το θέμα αυτό. ελπίζω να το και μπορώ να σας το πω ότι θα το παρακολουθούμε, αλλά επειδή αύριο θα ε, εγκριθεί σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ. Η συγγήτρια έχει και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ εκτιμώ τα σχόλιά σας και προσβλέπουμε στις διαβουλεύσεις με την Κομισιόν αύριο που πολλά συγκεκριμένα θα προσφέρει. Κυρία Γκέπχαρ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνούμε ε, στα περισσότερα που είπατε, εσείς και ο κύριος Παντσέρη. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να επικεντρωθούμε σε θέματα που μπορούμε να κάνουμε διαφορά σε κοινωνικό επίπεδο. Το θέμα των ενοικίων. Δεν λέω ότι δεν είναι πρόβλημα, αλλά λέω ότι δεν είμαι βέβαιη ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά ως κοινοβούλιο. Το ίδιο θα έλεγα και για τα φορολογικά κίνητρα. Μπορούμε να το δούμε λίγο μαζί αργότερα για να δούμε τι ακριβώς εννοείται. Ε, ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο που είπε ότι πρέπει να καθορίσουμε προτεραιότητες, να περιορίσουμε λίγο την, ε, το πεδίο. Εγώ προσπάθησα να το προσδιορίσω λίγο, το πεδίο που, στο οποίο πρέπει να εμβαθύνουμε και που θα πρέπει να αφορά την ΙΜΚΟ. Τώρα, για την ανάλυση επιπτώσεων, αντίκτυπο κλπ. Ε, πείτε μου τι ακριβώς εννοείτε, ποιοι τομείς θέλετε να ε, συμπεριληφθούν το θέμα ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς. Βέβαια ψηφίσαμε εδώ ε, την έκθεση Αρίας και δεν νομίζω ότι πρέπει να ξανανοίξουμε το θέμα αυτό. Ίσως μπορεί να παραπέμψουμε, αλλά δεν μπορούμε πάλι να μιλήσουμε για το ηλεκτρονικό εμπόριο που υπάρχει επίσης και στην οδηγία για τους καταναλωτές. Ο περιορισμός του ανταγωνισμού και αυτό το έθεσε ο Μάλκολμ Χάρμπορ και πράγματι θα πρέπει να το δούμε. Αφορά και το ζήτημα το, της διαφοράς τιμών και του κατακαιρματισμού. Τα ιδιωτικές ετικέτες ε, είναι καυτό θέμα και συζήτηση. Κάποιοι λένε ότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό για τον καταναλωτή, άλλοι λένε ότι περιορίζεται ο ανταγωνισμός. Οπότε οπωσδήποτε πρέπει να το δούμε και να κάνουμε μια συζήτηση που την καλωσορίζω. Η κυρία Ρούλ, να διευκρινίσω ότι όταν μιλώ για θέμητες εμπορικές πρακτικές εννοώ Β2Β β προς β. Ε, έχουμε οδηγία για το 2008 ή 6 για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές β, προς γ, δηλαδή επιχειρήσεις προς τον καταναλωτή. Β προς γ. Οπότε είναι επίμαχο και λεπτό θέμα η θέση, η κυρίαρχη η πρόσβαση για τους μικρούς, η πρόσβαση για τους ηλικιωμένους, πρόσβαση σε καταστήματα κοντά στο σπίτι τους, ώστε να μην χρειάζεται να πάνε με το αυτοκίνητο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να υπησέλθουμε πολύ σε τοπικού κανόνες ε, για την ίδρυση επιχειρήσεων, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μία πρόσβαση αυτό οπωσδήποτε θα πρέπει να το δούμε. Δηλαδή υπάρχει ανάγκη να εξασφαλιστεί η πρόσβαση. Η κοινωνική, ο κοινωνικός ρόλος και η λειτουργία των ε, καταστημάτων ως ε, τόπος ανθρώπινης επαφής για ηλικιωμένους, όπως είπε η κυρία Γκέμχαρτ, δεν ξέρω, είναι σημαντικό βέβαια, αλλά τι άλλο μπορούμε να κάνουμε αν όχι για να μιλήσουμε για την ε, ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη πρόσβαση. Για το χρονοδιάγραμμα έκανα πολλές διαβουλεύσεις πάνω σε αυτό το θέμα με τη γραμματεία γιατί οι εμπλεκόμενοι μου ζήτησαν να φροντίσω για ευρύτερες διαβουλεύσεις. Όλοι θέλετε να εργαστείτε επαγγελματικά και να είναι μια αξιόπιστη έκθεση, οπότε θα πρέπει να δούμε και όλες τις τροπολογίες σας. Αυτά που λέτε για τα σλότ, νομίζω ότι με την έκθεση ε, ζυβά γιατί το θεμητό και δίκαιο εμπόριο θα είμαστε εντάξει σε ό,τι αφορά με τις τρεις θέσεις, αυτά τα slots που ε, μας έχουν διατεθεί. Θα μπορούμε δηλαδή να ε, ε, ασχοληθούμε με την έκθεση αργότερα. Ας το δούμε όμως γιατί θα ήθελα να έχω το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή που πάει το Μάρτιο περίπου. Τώρα για το θέμα ουσίας, να πω στον κύριο Ροσφόρο ότι θα ήθελα να προτείνω αλλαγή τίτλου στην έκθεση γιατί δεν πρόκειται για το scoreboard, για αυτό τον πίνακα βαθμολογίας, ούτε για παρακολούθηση. Σίγουρα στηρίζεται σε αυτά που έχει χαρτογραφήσει ήδη η Κομισιόν Εκεί επάνω εντοπίζομαι προβλήματα, λύσεις και βέλτιστες πρακτικές, αλλά δεν περιοριζόμαστε σε απλή ανάλυση. Εμείς θέλουμε να προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις, οπότε η παρακολούθηση δεν είναι αρκετά θετική. Δεν με καλύπτει απόλυτα. Μπορούμε να δούμε τη λιανική αγορά, την αναζωγόνησή της, εντάσσεται στην, ε, στο μεγάλο ε, πυλώνα της εσωτερικής αγοράς, στο λιανεμπόριο είναι πυλώνας της εσωτερικής αγοράς, θα το δει η Επιτροπή και θα υποβάλει προτάσεις. Οπότε δεν είναι ε, μια έκθεση που περιορίζεται στην παρακολούθηση, αλλά είναι προσανατολισμένη προς τις λύσεις. Ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ συνεχίστε να υποβάλλετε σχόλια και παρεμβάσεις. Βεβαίως, πολύ σωστό, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, χρειαζόμαστε περισσότερο τομέα και για το σχέδιο επιχειρήσης προς ε, καταναλωτές, β' προς γ. Ε, περιμένουμε να δούμε και το κείμενο για την ε, νέα αγορά, οπότε εντάξει, θα το ξανασυζητήσω με το χρονοδιάγραμμα. Θα μιλήσω και με τον κύριο Χάρμπορ, γιατί μου έκανε την πρόταση τηλεφωνικά. Δεν παρευρέθη στη συζήτηση εκείνο σήμερα, οπότε θα τον ενημερώσω, όπως και εσείς θα του πω τι απόψεις υπάρχουν και κάποια καλή συμβαστική λύση θα βρούμε. Τώρα, κατεπηγόντως, να δούμε κάτι άλλο σήμερα. Το απόγευμα έχουμε μια πολύ σημαντική ακρόαση και ε, έχουμε πολλούς εθνικούς βουλευτές, 23 από 13 χώρες, 11 χώρες μέλη, 2 χώρες ΕΖΕΣ, Ελβετία, Νορβηγία, 18 υπαλλήλους από 13 κράτη-μέλη, και έχουμε συνολικά 41 εκπροσώπους εθνικών κοινοβουλίων και 4 ευρωβουλευτές. Ε, δεν θα ήταν τρομερό, ε, δεν θα ήταν ντροπή να είναι μόνο 3-4 ευρωβουλευτές εδώ. Οπότε ενημερώστε τις πολιτικές ομάδες ότι χρειάζεται προσέλευση καλύτερη. Εγώ θα ζητήσω συγγνώμη γιατί η Βελική Προεδρία ε, ανοήτως πώς και ειδικά σήμερα ε, διοργάνωσε την ε, εκδήλωση και ένα hearing για τις ε, δημόσιες υπηρεσίες και πρέπει να είμαι εκεί γιατί είμαι και στο Προεδρείο. Αλλά θα έρθω όσο γίνεται πιο γρήγορα. Φροντίστε παρακαλώ να μην είναι άδεια τα έδρανα το απόγευμα. Έτσι κι αλλιώς μπορούμε σήμερα το, πρωί να τελειώσουμε λίγο νωρίτερα με την έκκληση να έρθουμε το απόγευμα. Και, α, κόντεψα να το ξεχάσω. Μην ξεχνάτε ότι η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 8 Νοεμβρίου όπου θα ψηφίσουμε και την έκθεση του κυρίου Ζουβέν, πολύ σημαντικό, μην το ξεχάσετε. Βεβαίως θα λάβετε και πρόσκληση, αλλά υπενθυμίζω ότι η προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ είναι Δευτέρα 8 Νοεμβρίου. Και ε, διακόπτεται τη σε αυτό το σημείο αυτό.